Right, can I call the meeting to order? Να ξεκινήσουμε συνάδελφοι. Πρέπει να δώσουμε στο ένα το περισσότερο χρόνο στους συναδέλφους για τη συνεδρίασή μας. Υπάρχει την έγκριση στη μέση της διάταξης, αν συμφωνείτε. Εντάξει. Έχω μονάχα μία ανακοίνωση ως πρόεδρος. Η συνεδρίαση σε την προετοιμασία του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών στις 17 Οκτωβρίου, η οποία θα γινόταν η προπαρασκευαστική συνεδρίαση αύριο, τελικά χρειάστηκε να αναβληθεί. γιατί το αρμόδιο άτομο δεν μπορεί να είναι παρόν. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρία της 7ης Ιουλίου στο φακελό σας. Όπω λέει και ο κύριο Μπροκ, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει τώρα, από τώρα μέχρι το τέλο τη συνεδρία, θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στη συνάντηση με την Χέλγα. Είναι μεγάλη χαρά να είσαι εδώ ανάμεσά μας. Προφανώς δεν χρειάζεται να σε παρουσιάσω. Έχουμε παρακολουθήσει από πολύ κοντά το έργο σου στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ρόλο σου ως ε, Γενικής Γραμματέας, Γραμματέος. Είμαστε πάντα πολύ χαρούμενοι να μπορούμε να σε καλωσορίσουμε ως Γενικό Γραμματέα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και είναι και μια ευκαιρία για τους συναδέλφους να συζητήσουμε το θέμα του Αφγανιστάν και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα θελήσουν πιστεύω οι συνάδελφοι να συζητήσουμε. Η συνδιάσκεψη του Βρυξελών για το Αφγανιστάν έγινε στις 5 Οκτωβρίου. 75 χώρες ε, είχαν συμμετάσχει και έδωσαν μια κοινή δήλωση η οποία υπογραμμίζει την συλλογική τους δέσμευση να εντείνουν τη συνεργασία τους για να μπορέσει να έχει μια μεταμόρφωση του Αφγανιστάν σε μια κοινωνία με αυτονομία και ικανότητα διακυβέρνησης η Αντιπρόεδρος και είπα ότι εκπρόσωπος είπε ότι έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες της και σε ό,τι αφορά τα ποσά τα οποία υποσχέθηκαν οι δωρητές, 36 εκατομμύρια για τις προτεραιότητες Εθνική Ανάκτησης 13,6 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια τα οποία είναι υπέρ των προτεραιοτήτων του Αφγανιστάν. Και νομίζω ότι ένα από τα θέματα για τα οποία θέλουμε να ακούσουμε από σένα είναι οι συνέπειες της έκπνοης του προηγούμενου προγράμματος και εδώ θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί του Αφγανιστάν και ποιες είναι οι μελλοντικέ μας ε, προοπτικές για να δώσουμε συνέχεια στην αποστολή της ε, ΚΕΠΑ η οποία βρίσκεται στο Αφγανιστάν από το 2007. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Έχουμε μια χώρα η οποία βρέθηκε μέσα στη δίνη μιας από τις χειρότερες συγκρούσεις στον κόσμο και θέλουμε να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον για αυτή τη χώρα και περιμένουμε να ακούσουμε αυτά τα οποία θα μας πει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Τα εκτιμώ ιδιαίτερα. Να σας πω ξεκινώντας ότι η διάσκεψη ήταν μεγάλη επιτυχία και δεν ήταν κάτι εύκολο από την αρχή. Προηγήθηκε ένα έτος προπαρασκευαστικών εργασιών και από διδοεπένους τους συναδέλφους μου που έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είχαμε πάνω από 70 χώρες που συμμετείχαν, 26 διεθνούς οργανισμούς, και ε, παραπάνω από μισές από αυτές τις χώρες ήρθαν σε υπουργικό επίπεδο. Το ε, βαθμός αυτός ε, συμμετοχής σημειώνει την τεράστια επιτυχία. Μια άλλη πλευρά του διονομίσματο ήταν η διάσκεψη στη Βασοβία του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη των Αφγανικών δυνάμεων το 2016. Εμείς είδαμε την μη στρατιωτική πλευρά στη διάσκεψη. Είπατε εκπρόσωπος, όπως είπατε, ανέφερε ότι εκπληρώθηκαν όλε τι προσδοκίε. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τι υποσχέσει. γενικά υπάρχει κάποια κόποση των χορηγών γενικότερα, αλλά με τις προσωπικές προσπάθειες της ΥΠΑ της εκπροσώπου, πολλοί από τους εταίρους μας και πολλών από τους εταίρους μας και των δικών μου συναδέλφων καταφέραμε να μας υποσχεθούν 15,2 δισεκατομμύρια για αναπτυξιακή βοήθεια μεταξύ 2017 και 2020 για το Αφγανιστάν. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι επίσης ε, ε, σημαντικό γιατί δεν ήταν μόνο ε, η χρηματοδότηση θέμα, υπήρχε και μια πολιτική πτυχή. Οι γείτονες του Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Ινδία, η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν συμμετείχαν στη διάσκεψη. και παρατηρήθηκαν να, να ασκήσουν όποια επιρροή μπορούν για σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα. Οι προκλήσεις πριν από τη διάσκεψη, στο διάστημα δύο ετών ε, ε, με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ε, υπό τον πρόεδρο Απτούλα, ήταν να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση. Το ίδιο ήταν και η πρόκληση κατά τη διάσκεψη, κυρίως όσον αφορά την εκλογική και την συνταγματική μεταρρύθμιση. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να επικαιρώσουν τις νέες κινήσεις συνεργασίας. Να υπογράψω επίσης ότι η διάσκεψη έλαβε χώρα πάνω σε ένα υποβαθρό διαρκώς ε, ε, εντυνόμενης κατάστασης ε, προβλήματων ασφαλείας με τους Ταλιμπάν να επιτίδεται συνεχώς στην Κοντούς αλλά χωρίς να καταφέρουν να καταλάβουν την πόλη. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αφγανικής ε, κυβέρνησης και της ομάδας του κ. Χέγκ Ματιά που αποτελεί μήνυμα προς τις άλλες ένοπλες ομάδες ότι είναι δυνατή η διαπραγμάτευση λύσεων. Εμείς βοηθήσαμε να διευκολυνθεί η κατάσταση και τώρα επιβλέπουμε την αρρωγή και την υλοποίηση συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ε, δικαιωματών των γυναικών. Στοιχείο που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της διάσκεψης, υπήρξε μια ξεχωριστή συνεδρίαση, θα αναφερθώ σε αυτή πιο λεπτομερώς. Διάφορες πολιτικές προτεραιότητες υπήρξαν ε, που χαρακτήρισαν όλη τη διάσκεψη από την εναρκτήρια εκδήλωση μέχρι τις διμερείς δηλώσεις υπενθυμίστηκε η σταθερότητα της κυβέρνηση κυβέρνησης εθνικής ονότητας, πρόοδος με την εκλογική και συνταγματική μεταρρύθμιση, παρακολούθηση των εκλογών και συνεχής μεταρρυθμίσεις ε, ε, στον τομέα των διοικητικό του Αφγανιστάν και ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών. Ανέφερθηκε η κυρία Μογκερίνη και στις ε, οργανισμούς, στους οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών και τόνισε την ανάγκη να εξελιχθεί η διαφθόρα και να εξυγχρονιστεί η διοίκηση στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος. Αυτά τα είχαμε προετοιμάσει ήδη πριν από ένα χρόνο, όπου εγώ συμμετείχα στην Υπουργική Διάσκεψη ε, στην Ασιατική Υπουργική Διάσκεψη στην Ινδία, σε στενή συνεργασία με του Αμερικανού εταίρου. Είχαμε προετοιμάσει τότε τα βασικά στοιχεία για τη διάσκεψη και αναφέραμε την ανάγκη εκ νέου δέσμευση ε, από αφγανική πλευρά. Ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Εδώ επιτεύχθηκαν πολλά. Ένα άλλο σημείο πέραν των δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσει και των υποσχέσεων χρηματοδότησης ήταν η περιφερειακή διάσταση. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην περιφερειακή διάσταση. Έγινε μια μικρότερη ε, συνάντηση ε, με τη Φεντερίκα Μογκερίνη, αλλά και ο διαρθρωτικός διάλογος με το Πακιστάν και η υπουργική συνάντηση με τις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας και διάφορες άλλες διμερείς συναντήσεις. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε και χαιρόμαστε που έγινε πραγματικότητα, το βασικό αποτέλεσμα είναι μια κοινή περιφερειακή συνένεση, να γίνουν νέες προσπάθειες κατευνασμού των σειράξεων που δι, ανοίγει ένα νέο παράθυρο ελπίδας. Αποτελεί ένα περιθώριο για μια κοινή βάση για περιφερειακή πολιτική στήριξη για μια ειρηνευτική διαδικασία τη οποία θα ηγείται το ίδιο το Αφγανιστάν χωρίς αποκλεισμού βάσει των δημοκρατικών αρχών ε, και ε, με τήρηση του Αφγανικού Συντάγματος ε, ενώ όλοι κατανοούν ότι θα χρειαστούν διαπραγματεύσει με τους Ταλιμπάν βάσει αυτών των αρχών. Επίσης ζητήθηκε η μετανάστευση και οι δράσει για το μέλλον δεν αποτέλεσαν κομμάτι τη διάσκεψη. Υπήρξαν κάποιε. Ε, δηλώσει τον τύπο που δημιούργησαν κάποια σύγχυση. Αλλά η συμφωνία υπογράφηκε έγκαιρα για τη διάσκεψη. Να πω ότι η αρνητική εικόνα που έδωσαν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωση ήταν λάθος. Δεν τέθηκαν όροι για την παροχή αρρωγής. Είναι λάθος αυτό, αυτός ο χειρισμός. Αυτό που συνέβαινε ότι καθιερώθηκαν οι όροι συνεργασίας ε, με την αυγανική κυβέρνηση χωρίς να επηρεάζεται η των μεταναστών, επηρεάζονται οι πρόσφυγες που ζητούν άσυλο το οποίο έχει απορριφθεί. Κάτι άλλο σημαντικό εδώ, με τη βοήθεια των Αμερικανών συναδέλφων, όλοι οι σημαντικοί παλιότεροι δωρητές ε, συμπεριλαμβανομένες της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας επικύρωσαν τις δεσμεύσεις τους αλλά η διάσκεψη όμω σήμανε επίση και μια νέα δέσμευση μη παραδοσιακών χορηγών. Και αυτό ήταν ένα αντικειμενικό σκοπό από την αρχή, την οποία επιδιώκαμε για 12 μήνε. Και εδώ ε, λάβαμε υποσχέσει χορήγηση από την Ινδία, το Πακιστάν, η Ινδία ένα δισεκατομμύριο, μισό δισεκατομμύριο το Πακιστάν, 100 εκατομμύρια η Σαουδική Αραβία και είμαι περήφανο να πω εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών ότι ανταποκρίθηκαν στι προκλήσει να διατηρήσουν το σημερινό επίπεδο δέσμευση που ανέρχεται σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ετησίω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη καθιστώντας τους ε, τον μεγαλύτερο συμμετέχοντα στην αναπτυξιακή βοήθεια στο Αφγανιστάν. Κάτι τώρα να σας πω για τις παράπλευρες συναντήσεις που έλαβαν χώρα, ειδικότερα αυτή που αφορούσε τη χειραφέτηση των γυναικών. Πρόκειται για μια εκδήλωση όπου συμμετείχαν 450 άτομα συμπεριλαμβανομένου ε, του Προέδρου και της συζύγου του, του κ. Αμπτούλα, της είπα της εκπροσώπου, του Επιτρόπου Νίμιτσα, ε, με μεγάλη προβολή στον τύπο. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι έστειλα ένα χειρό και εκτός ε, της διάσκεψης. Εγώ συναντήθηκα με τον, τη δόκτωρα Χαμπίβα Σαράμπη που συμμετείχε με σημαντικό ρόλο στη διαπραγματεύση με το Ρενευτικό Συμβούλιο και ήταν και πρώην κυβερνήτης μιας ε, επαρχίας του Αφγανιστάν. Όσον αφορά τις γυναίκες, αυτή είναι μια από τις θετικές ιστορίες. Από, τις, από τους 90 εκατομμύρια φοιτητέ, ε, ε, ε, ένα μεγάλο ποσοστό είναι κορίτσια, πολλές χιλιάδες δικαστές, πάνω από το 50%, των, 50 των βουλευτών είναι ε, γυναίκες. Εγώ αξιοποίησα την άτυπη συνάντησή μου με κάποιες ε, από τις γυναίκες για να τους ρωτήσω τι περισσότερο μπορεί να γίνει για να υποστηρίξουμε τις γυναίκες, όχι μόνο για να τις προστατεύουμε, τις γυναίκες και τα κορίτσια, αλλά για να υποστηρίξουμε και τη χειραφέτησή τους. Και η απάντηση που έλαβα ήταν πολύ απλή, η παιδεία. Η παιδεία είναι το κλειδί. Παιδεία για τα κορίτσια και για τα αγόρια και για τους άνδρες. Και αυτό επικυρώνει ότι η προσέγγιση μας είναι η σωστή. Θα ξέρετε ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζεται στην υποστήριξη της περιφερειακής, α, αγροτικής ανάπτυξης, της υγείας και της παιδείας, ώστε να έρθουν τα εμπόδια. Για να γίνει αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να εστιαζόμαστε στη χειραφέτηση των γυναικών του Αφγανιστάν. Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε την πρόσβασή τους στην αγορά και στη χρηματοδότηση. Έχουμε πολλά παραδείγματα επιτυχή, αλλά η δέσμευση είναι μακροχρόνια. Νομίζω ότι ο Τζον Κέρι είχε πει, το είπε στην ομιλία του στην αρχή, επιτύχαμε πολλά, αλλά για να μείνουν όλα αυτά και για να επιτύχουμε και άλλα, θα χρειαστεί δέσμευση μακροχρόνια. Αυτό ήταν επίσης και ένα από τα μηνύματα αυτής της εκδήλωσης ε, στα οποία συμφώνησε ολόκληρη η διεθνή κοινότητα. Να πω επίση ότι δεν θα κάνουμε κανένα συμβασμό καμία παραχώρηση. Προβλέπονται διάφορα προγράμματα και αρρωγή που θα βασιστούν στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις τοπικές κοινότητες συντονισμένα και ταυτόχρονα οι γυναίκες θα πρέπει να αποκτούν ευκαιρίες αμερόλεπτα και ουδέτερα στις περιφερειακές και αστικές περιοχές σε ολόκληρη την επικράτεια του Αφγανιστάν. Άλλη εκδήλωση ήταν για την περιφερειακή οικονομική συνεργασία υψηλοί εκπρόσωποι από 10 οργανώσεις, 23 χώρες συνήλθαν. Ήταν και ο πρόεδρος Αμπτουλά, Υπουργή Εξωτερικών, αναπληρωτές Υπουργοί από την Περιφέρεια. Όλοι οι συμμετασχόντες τόνισαν ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των βασικών δωρητών, των περιφερειακών παικτών, των κυβερνήσεων. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες εδώ, αλλά οι βασικές προτεραιότητες ήταν έργα υποδομής, δημιουργία διαδρόμων ενεργειακών, σιδηροδρομικών, ψηφιακών, αλλά και ήπια υποδομή, επιχειρηματικά δίκτυα και τα παρόμοια επιχειρήσεις ε, που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον ε, είναι σημαντικές. Τέλος, Τώρα οπωσδήποτε θα παρακολουθήσουμε, θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή σε σχέση με τις δεσμεύσεις ε, στον τομέα γυναικών και κοριτσιών. Όμως ε, θέλω να παραθέσω τον ίδιο τον πρόεδρο που είπε στη διάσκεψη ότι τα πιο σημαντικά θέματα είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Είπε άμα δεν επιδείξουμε πολιτική, πολιτική βούληση στην πράξη, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, οι υποσχέσεις θα μείνουν υποσχέσεις. Και νομίζω ότι αυτό που είπε ε, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χέλγα θα ακούσουμε στους συναδέλφους τώρα. Μία ερώτηση. Ξέρουμε ότι ο αριθμός των Αφγανών προσφύγων που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται αριθμητικά. Ε, και αυτό είναι ένα θέμα ανησυχίας. Πολλοί δεν θέλουν ε, να ε, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα εδώ, αλλά στην πηγή τους και υπάρχουν αντιφάσεις σε ό,τι αφορά την ε, εξωτερική πολιτική ε, στην Αφρική ή το Αφγανιστάν. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να μας πει συγκεκριμένα τι ε, αντίχτυπο είχε η διάσκεψη των δωρητών στους αριθμούς των προσφύγων και αν θεωρείτε ότι μια τέτοια διάσκεψη μπορεί να καταπιαστεί και να λύσει προβλήματα επιτόπου. Ο κύριος ε, Κάν από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, ΕΛΚ δεν βλέπω. Ευχαριστώ. Ε, χαιρετίζω αυτά που είπατε. Έχω κάποιες ερωτήσεις για το Αφγανιστάν. Επίσης, ε, ε, ε χαιρετίζω και την ομάδα TR. αλλά το πρόβλημα είναι η Ταλιμπάν. Αν δεν βρεθεί λύση, βλέπουμε κλιμάκωση κάθε χρόνο. Η Ταλιμπάν είναι και μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στο Αφγανιστάν. Τι βήματα λοιπόν θα γίνουν για να αντιμετωπιστούν. Επίσης, είναι καλό που ακούμε για τις δωρεές στο μέλλον. Αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τις δωρεές είναι και η διαφθορά. Τι μέτρα λοιπόν λαμβάνονται ώστε να μπορέσει η αφγανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ίδια περιοχή. Είδαμε τις προηγούμενες 93 ημέρες ε, στην ειδική πλευρά του Κασμίρ ε, απαγόρευση της κυκλοφορίας πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν, δεκάδες χιλιάδες τραυματίστηκαν, πάνω από ένα ε, εκατομμύριο σφαίρες ρίχθηκαν στους αμάχους και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Και οι δύο χώρες έχουν πολεμήσει πολλές φορές μεταξύ τους. Ε, το, Αφγανι, το Αφγανικό οπωσδήποτε ε, είναι ένα ε, πρόσθετο πρόβλημα τι γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας ώστε να κινηθεί προς την ειρήνευση και την ευημερία. Και βέβαια πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα του Κασμίρ. Τέλος, ε, η Συρία, λίγο μακριά βέβαια, αλλά θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Τι γίνεται με τη βοήθεια και την προστασία των αμάχων. Η Πατή εκπρόσωπος μίλησε για συνεργασία με στον Γενικό Γραμματέα. Ε, θα μπορέσει έτσι να λυθεί το πρόβλημα της βοήθειας προς τη Συρία. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι θέλουμε η σημερινή συζήτηση, ζητήσαμε να εστιαστεί η σημερινή συζήτηση στο θέμα του Αφγανιστάν και οι γενικότερες ερωτήσεις πιστεύω θα γίνουν καλόδεκτες αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο Αφγανιστάν γιατί θα έχουμε και καιρό να συζητήσουμε τα άλλα θέματα σε άλλες ευκαιρίες. Ο κύριο Αυστρεβίτσιο είναι ο επικεφαλή τη αντιπροσωπεία με το Αφγανιστάν. Καλώ ήρθατε, σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Σύνοδο των Δωρητών για το Αφγανιστάν ήταν μια πραγματική επιτυχία. Στη διάσκεψη λοιπόν των Βρυξελών ήταν πολλέ οι χώρε οι οποίε συμμετέσχαν και ενεργά με στόχο να μπορέσουν να βοηθήσουν το Αφγανιστάν. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει, γιατί και εγώ είχα την, ε, το προνόμιο να μπορώ να με παρών σε αυτήν την ε, συνδιάσκεψη, είναι ότι υπάρχει μια αιρεσιμότητα για την οικονομική βοήθεια προς το Αφγανιστάν, που αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές. Και βέβαια αυτή η αιρεσιμότητα είναι κάπως διαφορετική από την προηγούμενη. Πώς λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αιρεσιμότητα, ώστε όπως ελέγχθη προηγουμένως, να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά και να εξασφαλίσουμε καλύτερη διακυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Και δεύτερον, ο κύριος Κέρι έκανε μια σαφή δήλωση για την περιφερειακή ε, διάσταση και την ε, επίπτωση των δράσεων χωρών όπως η Κίνα. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να δούμε μια καλύτερη περιφερειακή συνεργασία γιατί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών, των χωρών της περιφέρειας ήταν πολύ σημαντική και για το μέλλον του Αφγανιστάν. Ο κύριος Στάνο, PCR. Σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και η τελευταία σας εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής μας και γι' αυτό θα ήθελα εκ βάθους καρδίας και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων ανεξάρτητα από πολιτικές οικογένειες και πολιτικές τοποθετήσεις θέλω να σας εκφράσω τον σεβασμό που έχουμε για την συνεργασία που είχαμε μαζί σας όλο αυτόν τον καιρό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο επόμενο εγχείρημα το οποίο θα αναλάβετε. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την ύπατη εκπρόσωπο και εσάς ε, την ίδια για την επιτυχία αυτής της συνδιάσκεψης. Προφανώς η αντιμετώπιση της ε, διαφθοράς είναι το πιο σημαντικό θέμα για μας όταν μιλάμε για την ε, δόρηση βοήθειας προς το Αφγανιστάν, για την ασφάλεια των εργαζομένων στα θέματα βοήθειας προς το Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν και η μείωση των ροών μεταναστών ώστε να μπορέσουν να μείνουν εκεί και όχι να κάνουν το δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι στην Ευρώπη. Θέλω να δείξω όμω ένα διαφορετικό θέμα δεν είναι ακριβώς το μήνυμα το οποίο μπορεί να θεωρήσετε ότι αποτελεί. Αλλά θα ήθελα να ξέρω αν έγιναν συζητήσεις στην συνδιάσκεψη αυτή σε σχέση με το, με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από το Brexit. Πώς θα αλλάξει η συμμετοχή του στο πολυμερές πρόγραμμα χρηματοδότησης. Θα ήθελα να ξέρω παγκοσχάρι τι θα γίνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ότι είναι διακυβερνητικό μπορεί φυσικά να παραμείνει εκεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Και παραδοσιακά ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης έχει πάει σε προηγούμενες, σε πρώην χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Αν ε, αποσυρθούμε τελείως από, το, <clears throat> την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπάρξει ανακατεύθυνση των δωρεών προς, ε, παραδείγματος χάρη, αφρικανικές χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι έγινε στη διάσκεψη και τι ελέγχθη σε σχέση με την Βρετανική συνεισφορά. Εξετάστηκε καθόλου το θέμα αυτό είμαι κάπως προσωρινός πρόεδρος αλλά ίσως θα ήθελε η Γενική Γραμματέας να αναφερθεί στο θέμα της ενδεχόμενης αλλαγής της χρηματοδότησης με το Αφγανιστάν. Η κυρία Λοχπίτερ. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Στίβενς για την παρουσίαση που μας έκανε. Θα ήθελα να σας θέσω ένα θέμα σε αυτό, για αυτό το κοινό, για την κοινή πορεία προς τα εμπρός. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 80.000 Αφγανούς οι οποίοι ζήτησαν άσυλο και απορρίφθηκε η αίτησή τους και με τη βία κινδυνεύουν να επαναπατριστούν στο Αφγανιστάν. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν λαμβάνει κανείς υπόψη την κατάσταση ασφαλείας που επικρατεί στο Αφγανιστάν όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το 2016 μέχρι τώρα είχαμε 5.000 εθελοντικές επιστροφές που έχουν οικογένεια εκεί, έχουν συνθήκες να ε, επανέλθουν. Αλλά όταν εμείς απελάβουμε προς το Αφγανιστάν άτομα τα οποία δεν έχουν κάποιο οικογενειακό ή κοινωνικό ιστό να τους υποστηρίξει και είναι τόσο άσχημη και δύσκολη η κατάσταση ασφαλείας και το αναφέρετε εσείς, η περιοχή που ελέγχουν οι Ταλιμπάν έχει ενισχυθεί, έχει διευρυνθεί περισσότερο από ότι πριν από πέντε χρόνια και η ΚΕΣΤΖΕ, μια γερμανική υπηρεσία υποστήριξης προς, τους, προς το Αφγανιστάν, έχει αποσυρθεί γιατί είναι δύσκολο να, δια, να διατηρήσει συνθήκες ασφαλείας. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς στους πρόσφυγες ότι πρέπει να ξαναγυρίσουν σε μια τόσο δύσκολη περιοχή. Μήπως υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσατε να εξετάσετε. Ο ως από την ομάδα των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να μιλήσω για την ατζέντα που περιγράψατε και συγκεκριμένα από τους μηχανισμούς για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλές δραστηριότητες στη μετεκπαίδευση, την επιμόρφωση ε, με μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών. Έχουν αρχίσει τέτοιες διαδικασίες και τι σχεδιάζεται για τα επόμενα χρόνια. Γιατί στο Αφγανιστάν αυτό είναι σημαντικός μοχλός για το μετασχηματισμό της κοινωνίας συμμετοχή γυναικών και νέων ανθρώπων βέβαια, ε, που θα αλλάξει ε, την κοινωνία και θα την κάνει πιο ανεκτική. Ευχαριστώ κύριο Σάλβια την ομάδα των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Και εγώ, ε, Ρίτσαρντ, θέλω να δώσω τις καλύτερες ευχές μου για το επαγγελματικό και προσωπικό σας μέλλον. Ήταν μεγάλη μου χαρά που συνεργάστηκα μαζί σας τα προηγούμενα χρόνια. Εύχομαι ότι καλύτερο. Μία ερώτηση σχετικά με το κατεμέ βασικό θέμα στο Αφγανιστάν. Όταν συζητούσαμε για το Αφγανιστάν πριν από λίγα χρόνια, θυμάμαι ότι η ιδέα ήταν να αποσυρθεί να, να, μείνει ο στρατός μέχρι το 2011. Και δεν έγινε αυτό λόγω της ισχύω των Ταλιμπάν, οι οποίοι α, ισχυροποιήθηκαν αντί να εξαφανιστούν όπως ελπίζαμε. Δεν εξαφανίστηκαν. Και ρωτώ, έχουμε δυνατότητα ανάληψης κάποιας πρωτοβουλίας ε, προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης στη χώρα αυτή γιατί είναι κάτι παραπάνω από προφανές για μένα ότι επειδή η σύγκρουση στο Αφγανιστάν δημιουργήθηκε από τον εξωτερικό παράγοντα, πρώτα από τη Ρωσία και μετά τους φίλους μας, τους Αμερικανούς και άλλους, ο μόνος τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι οι Αφγανοί να προσπαθήσουν να λύσουν μεταξύ τους με δραστήριο τρόπο τα προβλήματά τους. και εκεί ίσως θα μπορούσε να παίξει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα μου κάνανε εντύπωση τα λόγια του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν είπε ότι χρειαζόμαστε Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιος που θα συμμετέχει στις συζητήσεις γύρω από ένα τραπέζι όταν είναι περίπλοκα τα θέματα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν ε, θα συμβεί αυτό κατά από αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία εκεί όπου έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, όπου έχουμε ειδικό βάρος, ούτω ώστε να διευκολύνουμε τον διάλογο στο Αφγανιστάν. Μπορεί αυτός να είναι ένας καλός και σωστός ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κουκκίν για το έλκο. Ευχαριστώ Ρίτσαρντ. Καλό που σας βλέπουμε στο Προεδρείο. Βλέπω ότι εκτιμήθηκαν τόσα καράτη για αυτή την Επιτροπή μετά από πολλά χρόνια αφουσίωσης. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για το μέλλον. Και ελπίζω να σας ακούμε όλο και περισσότερο και το εννοώ θετικά. Κυρία Γενική Γραμματέα, Έχω μια πολύ γενική ερώτηση. Κάπου πριν από 10 χρόνια περίπου όλοι έλεγαν το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να χάσει το Αφγανιστάν. Δεν μπορεί να χάσει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Είναι το τελευταίο περιθώριο που μας μένει. Πώς θα σχολιάζετε αυτές τις δηλώσεις σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι για τα πολύ ευγενικά σας ε, λόγια κύριε Τάνοκ, ε, κύριε Κοκάν, κύριε Βάγκλ. Αλλά εδώ συζητάμε το Αφγανιστάν πολύ σημαντικό θέμα, οπότε δίνω το λόγο στην Γενική Γραμματέα. Um, uh, Ευχαριστώ. Να αρχίσω με τους ε, μετανάστες, πώς θα προχωρήσουμε ε, τις ε, λανθασμένες απόψεις που υπάρχουν. Όπως είπα, υπήρξε, υπήρξαν παραπλανητικές εκθέσεις είναι σαφές ε, ότι ο κοινός δρόμος μπροστά είναι κοινή δέσμευση που αναλάβαμε με την Αφγανική κυβέρνηση για να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση παράνομης μετανάστευσης. Πρόκειται και για το λαθρεμπόριο και για τη διακίνηση ανθρώπων ή διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής ε, Αφγανών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να μείνουν. Υπάρχουν κάποιες αρχές δηλαδή που ισχύουν, ε, αρχές ε, διεθνούς ε, δικαίου, η αρχή της μη επαναπροώθησης, άνθρωποι που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες προφανώς χρήζουν προστασίας. Αν δείτε και το ποσοστό αποδοχής των ετούντων άσυλο έχει αυξηθεί σε, κατά 60% κατά μέσον όρο που αναφέρεται σε αυτό που είπε η κυρία Λόχμπίλερ. Επίσης δεν υπάρχει αιρεσιμότητα και εδώ υπήρξε παραπλάνηση και είπα ότι εκπρόσωπος στην, ε, στις δηλώσεις της παρυφές ε, ε, της διάσκεψης το ξεκαθάρισε αυτό. δεν υπάρχει αιρεσιμότητα σε σχέση με την επιστροφή παράνομων μεταναστών. Υπάρχει Έγινε και μια ερώτηση για την ερεσιμότητα σχετικά με τις γυναίκες και την οικονομική βοήθεια. Και εδώ να απαντήσω άμεσα. Και εδώ δεν υπάρχει αιρεσιμότητα. Βέβαια, όταν πρόκειται για το πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα, εκεί θα παρακολουθήσω με εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής ατζέντα. Και άλλη ερώτηση έγινε εδώ, έγιναν πολλά. Οι Υπουργοί Οικονομικών προσεκλήθησαν να έρθουν στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός ε, ήρθε στις Βρυξέλλες, έγιναν καλές συζητήσεις ε, πολλοί διεφθαρμένοι δικαστές ε, απολύθηκαν για παράδειγμα. Η κυβέρνηση δηλαδή πολύ συγκεκριμένα προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Εμείς τους στηρίζουμε με τα διοικητικά μέτρα που και τη διοικητική βοήθεια που μπορούμε να λάβουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό πέρα από την υποστήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου, ε, την εκπαίδευση και την υγεία. Άλλη ερώτηση αφορούσε την Ινδία και το Πακιστάν. Είναι πολύ ευαίσθητα τα θέματα αυτά, το ξέρετε. Ε, συνεχώς τα συζητούμε στο διάλογο και με τις δύο χώρες ε, σε επίπεδο είπα της εκπροσώπου και στο δικό μου το επίπεδο και σε άλλα επίπεδα και ήταν κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου με το Πακιστάν. Ε, έγιναν όλα, όλες αυτές οι συζητήσεις όπως και με τον Ινδό Υπουργό Εξωτερικών οι γυναίκες και τι κάνουν αν κατάλαβα καλά, για να ε, προωθήσουμε την εκπαίδευση, κατάρτιση γυναικών και πώς τις εντάσσουμε περισσότερο. Εδώ το βασικό είναι η εκπαίδευση. Εδώ έχουν γίνει πολλά. Και αυτό το θέμα το συζήτησα και με τις γυναίκες που συμμετείχαν για να δούμε είμαστε στο σωστό δρόμο, τι μπορεί να γίνει. Και προς έκπληξη μου ε, άκουσα τις γυναίκες να λένε ότι πρέπει να δεχτείτε την πραγματικότητα μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας και πρέπει να μας βοηθήσετε με την εκπαίδευση ε, υπό την ευρία έννοια της. Παιδεία για όλους. Βέβαια προσφέρουμε κατάρτιση για τις γυναίκες, υπάρχουν προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί και στους κόλπους της Ένωσης. Ε, προωθούμε ευκαιρίες ε, στα διαδρομίες για τις γυναίκες και στο Business Forum. Υπήρχαν και άλλα business φόρα, τα οποία ειδικά αποσκοπούν στο να βοηθήσουν την ε, πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση και στον επιχειρηματικό κόσμο. Άλλη ερώτηση αφορούσε την ε, νοσιακή χρηματοδότηση και τι προοπτικές έχει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω γιατί δεν συζητήθηκε στη διάσκεψη, αν και το θέμα βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Ε, η ερώτηση του κ. Βάιγκλ για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ήδη πάρα πολύ ενεργά. Η υπατή εκπρόσωπος ε, έπαιξε ρόλο διευκολυντικό για την ειρηνευτική ε, συμφωνία ε, με την ομάδα που δεν είναι που δεν είναι πολύ η μεγαλύτερη ομάδα αλλά ήταν ισχυρό το μήνυμα που δόθηκε σε άλλες ομάδες και στους Ταλιμπάν. Το σημαντικό είναι ότι αυτά που συμφωνήθηκαν θα υλοποιηθούν και είναι και βιώσιμα. Και έτσι αποστέλλεται και στην κυβερνητική πλευρά ένα μήνυμα. Τώρα εξετάζομαι τι, τρόπους υπάρχουν, τι τρόποι υπάρχουν για να ε, εφαρμοστούν τα μέτρα. Ε, εδώ και ο ρόλος των γυναικών είναι σημαντικός και το τόνισαν. Ο κύριος Κούκαν για τον ΝΑΤΟ που δεν μπορεί να χάσει το Αφγανιστάν. Εγώ θα έλεγα ότι εμείς δεν μπορούμε να χάσουμε το Αφγανιστάν. Γιατί δεν είναι μόνο θέματα ασφαλείας για μας ε, στα, ιστορικό πλαίσιο μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Είναι και πολιτικό θέμα, είναι και ανθρωπιστικό θέμα. Γι' αυτό μένουμε ε, ενταγμένοι. Είναι και σημαντικό το Αφγανιστάν για το περιφερειακό πλαίσιο. Η εστίαση αυτής της διάσκεψης ήταν κυρίως στο Αφγανιστάν. Αλλά τους προηγούμενους μήνες, χρόνια μπορώ να πω, προωθούμε και περιφερειακή διασυνοριακή προσέγγιση. Δεν ήταν τυχαία η συνάντηση με τις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας συζητήθηκε πολύ η διασυνοριακή συνεργασία. Έχουμε και τον διάλογο για την ασφάλεια που γίνεται μια φορά το χρόνο με τις πέντε χώρες κεντρικής αστείας που προσπαθούμε να προωθήσουμε ένα θετικό αφήγημα και για τη συνεργασία και για οικονομικά θέματα. Είναι η λιγότερο ολοκληρωμένη περιφέρεια του κόσμου αυτή. Υπάρχει δηλαδή πολύ ε, ε, δυναμικό που δεν έχει αξιοποιηθεί και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Και το θέμα της συνδεσιμότητας είναι σημαντικό. Ε, υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ που χρηματοδοτεί η Κομισιόν και βοηθούν την περιοχή και έχουν όλα αυτά σημασία που ξεπερνούν το ίδιο το Αφγανιστάν. Είναι πολύ πιο σημαντικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά, πιστεύω, από τότε που έχετε έρθει ενώπιον της Επιτροπής μας που συζητούμε το θέμα αυτό. Θέλω να σας ε, ευχαριστώ για τη συμβολή σας και πιστεύω ότι θα έχουμε και στο μέλλον ευκαιρίες να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Τώρα, ο κύριος Μπρόκ είναι ο εισηγητής για τις ε, εκθέσεις για την ΚΕΠΑ που είναι τα θέματα που ακολουθούν για το, την συμφωνία μεταξύ Κολομβία, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολομβίας και Εκουαδόρ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι να έρθει λοιπόν ο κύριος Μπρόκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Φαν Μπάρεν, ο σύντροφος Φαν Μπάρεν θα ήθελε να λάβει το λόγο. Όχι, αργότερα. Καλώς ήλθατε για το σημείο 5 της σημερινής διάταξης. Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Έχετε ενώπιον σας την έκθεση, το σχέδιο έκθεσης. Δεν θέλω τώρα να σας το παρουσιάσω εν λεπτομερία. Θεωρώ δεδομένο το έχετε διαβάσει όλοι προσεκτικά. Κάποιες εισαγωγικές μονάχα παρατηρήσεις θα ήθελα να θέσω. Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. 8 Νοεμβρίου θα γίνει συζήτηση στην Επιτροπή μας μαζί με τους ε, εθνικούς κοινοβουλευτικούς και αυτό μπορεί να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση να ακούσουμε τις απόψεις και των συναδέλφων που είναι εθνικοί. Στις 15 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε λοιπόν για το θέμα αυτό και θα έρθει στη συνέχεια στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο κανονικά. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις που έχουν γίνει στην ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις ή τουλάχιστον είναι πιο σαφείς και έντονες από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αν δεν είναι πιο μεγάλες. Προφανώς η εκθεσία ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά ασχολείται και με την συνολική στρατηγική της ε, του είπα της εκπροσώπου και αυτά τα οποία διαμήθησαν στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στην Βρατισλάβα. Υπάρχει και μία σειρά από εθνικές πρωτοβουλίες όπως είναι η γαλλογερμανική πρωτοβουλία, υπάρχει η ομιλία του Jean-Claude στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως είπα η στρατηγική της Μπρατισλάβα. Ο, ο δικός χάρτης που προήλθε από τη συνάντηση της Μπρατισλάβα την, το Δεκέμβριο θα έρθει στο, στην ημέρησια διάταξη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το θέμα αυτό και είναι πολύ καλό ότι θα το έχουμε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί ως τμήμα της στρατηγικής Πατσισλάβας το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο θα πρέπει το Δεκέμβριο να επιληφθεί πιο συγκεκριμένα για το θέμα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι η χρονική αλληλουχία για αυτήν την έκθεση θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε και κάποιες προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ασχολείται επίσης η έκθεση με την ε, ε, γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν φαίνεται ιδιαίτερα λαμπρή αυτή τη στιγμή και με τα συμπεράσματα τα οποία εμείς θα πρέπει να αντλήσουμε από τις εξελίξεις που έχουν λάβει η χώρα στις ε, χώρες της περιοχής, όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και την Λευκορωσία και άλλες. Και φυσικά πρέπει να υπάρξει και μια συζήτηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Πιστεύω, εδώ και δέκα μέρες τουλάχιστον πιστεύω, ότι αυτή η συζήτηση και σε σχέση με τη Ρωσία είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συζήτηση για την ανατολική μας γειτονία. Και έχω λοιπόν καταβάλει μία προσπάθεια. Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα πολλαπλά ερωτήματα στα οποία περιλαμβάνεται και η συνεργασία με τη Ρωσία για επιληθούν διεθνείς κρίσεις, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε θέματα όπως ε, με την Ουκρανία που έχουν οδηγήσει σε παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με τη Ρωσία παρά όλα αυτά τα οποία γίνονται λόγω της Ουκρανίας. Από τότε που η Ρωσία δεν είναι πια εταίρος για μια ελληνική επίλυση της ε, σύγκρουσης στη Συρία, αλλά έχει εμπλακεί ως ένας από τους αντιμαχόμενους, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση, κάτι το οποίο σημαίνει πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Παραδείγματος χάρη, πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τις ε, τις κυρώσεις οι οποίες ουσιαστικά κρατάνε για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά τις ξεχνάμε. Πηγαίνουν πολλοί πολιτικοί από τη Γερμανία και άλλες χώρες στη Ρωσία. Νομίζω ότι έχει κάθε νόημα να έχουμε ε, ανανέωση των κυρώσεων όχι κάθε έξι μήνες αλλά κάθε ένα χρόνο ώστε να γίνει σαφές ότι το εννοούμε και δεν είναι απλώς κάτι το οποίο αλλάζει κάθε έξι μήνες. Πρέπει όμως να σκεφτούμε και επίσης σε ό,τι αφορά το καθεστώς των κυρώσεων αν θα πρέπει σε σχέση με την απαγόρευση εξι, ε, εξαγωγών να περιλάβουμε και προϊόντα υψηλή τεχνολογία, τα οποία έχουν να κάνουν με του υπολογιστέ, με προϊόντα υψηλή τεχνολογία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε, σε οπλικά συστήματα κτλ. πρέπει να περιληφθούν όλα αυτά στο εμπάργο, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται όπλα από τη Ρωσία για να βομβαρδιστούν μέχρι και νοσοκομεία. Και ένα ευρύτερο θέμα είναι πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε τι καλύτερε συνθήκε για την κοινή αυτή πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις πολέμου και τρομοκρατίας. Πολλές φορές συνδέονται τα δύο φαινόμενα μεταξύ τους. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα και φυσικά και τις ρίζες <clears throat> του μεταναστευτικού προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο προσεκτικά τη σύνδεση το, της ΚΕΠΑ με εμπορικές συμφωνίες και άλλα τέτοια συναφή ζητήματα. Και αυτό σίγουρα έχει σημασία σε ό,τι αφορά την Αφρική. Το γεγονό ότι οι άνθρωποι στην Αφρική δεν έχουν καμία προοπτική, το γεγονό ότι υπάρχει μια τεράστια δημογραφική αύξηση του πληθυσμού στην Αφρική, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο τη συζήτηση για την ε, αντιμετώπιση των μεσταυτικών ροών όλα αυτά που κάνουμε σε ό,τι αφορά την κατανομή σε ποσοστό των ε, προσφύγων, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, η συμφωνία με την Τουρκία, η προσπάθεια αντιμετώπισης των διακινητών, όλα αυτά είναι ένας αγώνας κατά των συμπτωμάτων, αλλά όχι κατά της ε, πραγματικής αιτίας. Στην Αφρική θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανάπτυξης και αυτό είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πιο πολυσχηδή ε, εξωτερική πολιτική που λαμβάνει υπόψη θέματα εμπορικών συμφώνιων, κλιματικής αλλαγής και τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε μια καλύτερα διαμορφωμένη εξωτερική πολιτική η οποία θα είναι σε θέση να επιλύσει τα προβλήματά μας και που δεν θα έχει σαν στόχο μονάχα να θωρακίσει την Ευρώπη από μεταναστευτικές ροές. Για να μπορούμε να μην έχουμε υψηλό αριθμό μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη, πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εξωτερική πολιτική, μια καλύτερη εμπορική πολιτική, μια καλύτερη αναπτυξιακή πολιτική. Και επομένως, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της ε, συζήτησης. Πρέπει να συζητήσουμε προφανώς και τις πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων και την, ε, τον οδικό χάρτη της ε, Βρατισλάβας. Αλλά όλα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν και σε πιο έντονη συνεργασία, παραγωγός χάρη στον τομέα των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά την ε, δημιουργία μονίμων δομών άμυνας και συνεργασίας, την υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού φορέα για την άμυνα και την προμήθεια οπλικών συστημάτων, όλα αυτά τα θέματα τα οποία πριν από έξι μήνες δεν τολμούσαμε να τα προφέρουμε γιατί δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα και να προκαλέσουμε ένα ενδεχόμενο Brexit, τότε ενδεχόμενο, τώρα πραγματικό. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα τώρα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και όλα τα κράτη-μέλη κινούνται πια προς αυτή την κατεύθυνση. και που Αντίθετα από τον Υπουργό Εξωτερικών της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Υπουργό Άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου τα κατανοεί καλύτερα. Αυτή τη στιγμή ο Υπουργό Άμυνα τη Μεγάλη Βρετανία είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά γιατί αυτά οδηγούν σε προβλήματα στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας είπε όλα αυτά μας βοηθάνε ως ΝΑΤΟ. Και πιστεύω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα τονίσουμε και να πούμε στους Βρετανούς συναδέλφους ότι εάν αυτοί θέλουν να φύγουν, δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα μας πούν τι θα κάνουμε στον αμυντικό τομέα. Θέλουμε για τον Brexit να κρατήσουμε μια επικοδομητική στάση για να διαφυλάξουμε και τα κοινά συμφέροντα, αλλά Πρέπει να υπάρξει fair game, δίκαιη αντιμετώπιση από όλες τις ε, πλευρές, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα πέρα από αυτά να ακούσω και τις δικές σας ε, προτάσεις, τις δικές σας συστάσεις και είμαι πάντα έτοιμος να συζητήσω οποιαδήποτε από τις προστάσεις αυτές και είμαι έτοιμος να δεχθώ τις δικές σας συνεισφορές για να επιπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ποιος έχει το λόγο. Η κυρία Κανιέτη. Ευχαριστώ. Δεν περίμενα να είμαι η πρωτόκλητη. Κύριε Πρόεδρε, να πω καταρχήν ότι χαίρομαι για την έκθεσή σας γιατί ακριβώς πιάνει την σημερινή δυναμική. Θέλω να σχολιάσω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, είναι καλό που καλείται τα κρατη με να δεσμεύσουν το 2% του εγχωρίου προϊόντος στην άμυνα και 20% του αμυντικού προϋπολογισμού σε μεγάλους εξοπλισμούς αμυντικούς. Επίσης, θα έλεγα ότι παρόμοια δέσμευση ε, για τη διπλωματία άμυνα ανάπτυξη θα πρέπει να καλύπτονται με το 3% του καθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Τώρα, για την κεντρική διοίκηση. Ε, από τότε που άρχισε να γίνεται αυτή η συζήτηση για την κεντρική διοίκηση, Είχα, έκανα διαβουλεύσεις και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με το Υπουργείο Άμυνας στη Λετωνία και η έννοια αυτή, headquarters, κεντρική διοίκηση, δύσκολα γίνεται αποδεκτή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για τη δημιουργία νέας δομής για να αυξηθεί ο αριθμό των στρατηγών, όπως μου είπε κάποιος σύμβουλος. Όχι. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε δυνατότητες σχεδιασμού, πολιτικού σχεδιασμού, για να συντονίζουμε καλύτερα ε, ε, υποδομές στρατιωτικές και μη στρατιωτικές. Ευχαριστώ και θα ε, υποβάλω, όπως καταλαβαίνετε, τις σχετικές ε, τροπολογίες ε, στην εκθέσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα διαβάσω αυτό που έγραψε ο Σχιώδης ο εισηγητής. Ο κύριος Φλέγκενστάιν. Πράγματι μπορεί. Λοιπόν, να δούμε τι έγραψε Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον πρόεδρο της ΑΦΕΤ ε, Αλμαρ Μπρόκ για το σχέδιο έκθεσης το οποίο λαμβάνει υπόψη τη νέα παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου και συζητήθηκε από την Επιτροπή μας στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 6 Ιουλίου. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις και οι πολίτες της Ευρώπης έχουν προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο αποτελεσματική από τη σήμερα. Επίσης αναμένουν να προστατεύει τις ζωές τους, το επίπεδο διαβίωσής τους, να προωθεί αξίες όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την αλληλεγγύη και τη διεθνή συνεργασία, την πολιτική και οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια στην άμεση γειτονία και να συμβάλλει ε, αποτελεσματικά σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ε, της τρομοκρατίας και άλλων προκλήσεων. Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι σημαντική η τακτική αναθεώρηση και αν χρειαστεί ανασχεδίαση της παγκόσμιας στρατηγικής. Προτείνουμε λοιπόν μια αιτήσια συζήτηση για την ε, τρέχουσα κατάσταση και το καθεστώς υλοποίησης αυτή η νέα στρατηγική και νέες πρωτοβουλίες ενίσχυσης ε, ε, της παγκόσμιας στρατηγικής για την ασφάλεια ε, θα συμπεριλάβουν και αυτή την έκθεση ω στοιχείο τους και θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις συνθήκες που υπάρχουν. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα να παράσχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινότητας ασφάλειας με την απόκτηση όχι μόνο περισσότερων όπλων, αλλά αποφεύγοντας τον κατακαιρματισμό των πόρων των κρατών μελών και βελτιστοποιώντας αυτούς τους πόρους μέσω της εντονότερης και εντατικότερης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Αλλά θεωρούμε ότι η δύναμη της ευρωπαϊκής διπλωματίας, όπως λέει και ο εισηγητής, θα πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και της πολυμερούς διπλωματίας η κοινή πολιτική ασφαλεία και αμυντική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει πιο αποτελεσματικέ τι επαφέ μεταξύ κυβερνήσεων και έτσι είναι σημαντικό να απογειώσουμε την, την υπηρεσία Ευρωπαϊκή Εξωτερικής δράση και τι ε, δυνατότητες στρατηγικού σχεδιασμού τη με σημαντική ευρωπαϊκή συνιστόση. Υποστηρίζουμε τι σχετικέ συστάσει στο σχέδιο έκθεση. Αυτά λέει ο σχέδιο συζητητή συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να πω προσωπικά, στο Κοινοβούλιο έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να εντείνουμε την έρευνα και ανάπτυξη για την άμυνα και να παρατηρούμε τα κρατημέλη προς την ίδια κατεύθυνση. Αλλά θεωρώ ότι και τα ζητήματα του εμπορίου που και εσεί ε, και στο πλαίσιο αυτό οι, οι συμφωνίες ε, ε, εξοπλισμού θα πρέπει να γίνονται με τρόπο συνεκτικό ώστε τα κράτη-μέλη να πραγματοποιούν τις εξαγωγές ε, όπλων και τις συμφωνίες εξαγωγής όπλων ως εργαλεία εξωτερικής πολιτικής. Να υπάρχει κάποια εναρμόνιση δηλαδή σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τόσο πολλά προβλήματα στη δική μας Ήπειρο και δεν λέω ότι η Λατινική Αμερική δεν είναι σημαντική, το ίδιο και η Αφρική, το ίδιο και η Ασία. Αλλά εδώ γύρω έχουμε τόσα πολλά προβλήματα στην περιοχή μας και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε στην έκθεση ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τις δικές μας αμυντικές δυνατότητες. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα χρήματά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον πιο αποτελεσματικό αλλά πρέπει να συζητήσουμε και για το τι γίνεται με το ΝΑΤΟ, το οποίο θα είναι ζωτική σημασία και θα γίνει ακόμη σημαντικότερο καθώ η Βρετανία πρόκειται να καταλήψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη Ρωσία, η προσέγγιση δύο οδών που προτείνεται, η συνομιλία με την κοινωνία των πολιτών και οι κυρώσεις. Και μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν έχει κάνει τίποτα που να οδηγήσει σε μετριασμό ή σε απόσυρση των κυρώσεων. Και δεδομένου ότι δυνάμεις πυροβολικού από τη ρωσιακή επικράτεια μετέβησαν ε, στην περιοχή που όπου βρίσκονται οι αντάρτες στην Ουκρανία και μετά επέστρεψαν στη Ρωσία θα μας δώσει όλο και περισσότερες πληροφορίες για την εμπλοκή της Ρωσίας και ίσως να απαιτηθούν περισσότερες κυρώσεις αντί για λιγότερες, αλλά θα το δούμε. Εγκρίνουμε την έκθεσή σας, θεωρούμε την εξαιρετική επί της ουσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Συμφωνούμε με τα περισσότερα από όσα λέτε και ειδικότερα όσον αφορά την παγκόσμια αξιολόγηση των βασικών αιτιών, των μεγαλύτερων κρίσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική αυτή τη στιγμή. Κάποια πράγματα μας ε, ανησυχούν, θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες, απλά να τονίσω δύο. Πρώτον, θεωρούμε ότι η εικόνα δεν είναι τόσο απεσιόδοξη όσο την απεικονίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά δεν είναι πολύ καλή στην αυτοπροβολή της στους ίδιους πολίτες της. Ε, ξέρετε και η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία έχει κάποιες επιτυχίες που ε, ελάχιστα γίνονται γνωστέ εκτός. Οπότε δεν είναι όλα μια αποτυχία. Συμφωνούμε απόλυτα ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να εντοχθεί πλήρε ε, ε, στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία και στην αμυντική πολιτική και ότι η εξωτερική μα ανεπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να μα καθοδηγεί στη γενικότερη αξιολόγησή μα των προτεραιοτήτων. Αυτό που μα ανησυχεί είναι ε, ότι γίνεται μεσοπρόθεσμα με τις μεταναστευτικέ ροέ πώς θα δρομολογήσουμε πόρους ε, ε, λέμε προς ε, τις σχετικές περιοχές και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε την πρόληψη των σειράξεων. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την επίληξη των σειράξεων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική σε ορισμένες περιοχές από ότι η άμεση εμπλοκή. θα υποβάλουμε τις σχετικές τροπολογίες και υποστηρίζουμε γενικά την έκθεση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα με αυτή την έκθεση. Παρά είναι καλή και δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να την βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πιστική και ρεαλιστική, αλλά όχι η τοπαθή αξιολόγηση της διεθνούς κατάστασης και υπάρχει μια νέα πραγματικότητα που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Ωστόσο, πολύ υπευθύνοι ε, αποφάσεων ε, και ε, όσοι ηγούνται της κοινή γνώμης προτιμούν να μένουν στο χθε, ε, πιστεύοντας ότι θα αποκατασταθεί αυτό το χθε. Αυτή η έκθεση απεικονίζει μια νέα πραγματικότητα και καθιστά σαφές ότι οι νέε κρίσει αποτελούν μια ευκαιρία, είναι μια θετική νότα αυτή, όχι το παθή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο παγκοσμίω, εφόσον τα κράτη-μέλη μιλούν με μία φωνή και δρούν από κοινού. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά αυτό θα σήμαινε πρώτα απ' όλα η οικονομική συμβολή, η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Διαφωνώ λίγο με την παράγραφο 8, όπου η συγγετή συμπεραίνει ότι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων σε εποχές δημοσιονομικών περιορισμών είναι να αυξηθούν οι συνεργασίες, εντείνοντας την αμυντική συνεργασία. Δίκιο έχετε εμένα, αλλά το ερώτημα είναι πότε θα έρθει η στιγμή που δεν θα υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί. Πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή νοοτροπία. Διότι αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε επαρκώς σε εποχές κρίσης, τι θα κάνουμε αύριο αν επέλθει πόλεμος. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η χρηματική συμβολή όλων για την άμυνά μας θα προστατεύσει όλους μας στο μέλλον. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποστηρίξουμε να υποστηρίξουν όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου την παραγραφό 9. Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα ότι απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη και να χρησιμοποιηθεί η, η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου έχοντας αυτό στο νου μας. και πιστεύω αναφέρεται πολύ σωστά αυτή τη μόνιμη δομή συνεργασίας που προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνα. Τώρα όσον αφορά την υλοποίηση. Η κοινή χρήση των μυστικών πληροφοριών με τη Europol και τη Eurojust αναφέρεται εδώ, αλλά πιστεύω ότι πιο συγκεκριμένα πρέπει να επισημάνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Στη διασκέψη της Κρακοβίας την περασμένη εβδομάδα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αναφέρθηκε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών λειτουργεί μεταξύ των κρατών μελών εφόσον υπάρχουν καλές προσωπικές σχέσεις μεταξύ των αντίστοιχων αξιωματούχων, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτόματη. Τώρα όσον αφορά τη Ρωσία, συμφωνώ απόλυτα με την έκκληση προς μια πιο ρεαλιστική στρατηγική δεν έχουμε περιθώριο να ε, είμαστε κατακαιρματισμένοι. Τα αποτελέσματα που θα φέρουμε με τη Ρωσία θα βασιστούν στη δική μας συνεργασία. Αντί να διστάζουμε για το κατά πόσο θα λάβουμε περαιτέρω κυρώσεις ή όχι. Και μετά στην παράγραφο 19 ε, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το κείμενο πιστεύω, να εμβαθύνουμε τη σχέση με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά είναι κάτι που όχι μόνο εξυπηρετεί τα στρατηγικά μας ε, συμφέροντα, αλλά ε, είναι κάτι που θα βοηθήσει τις, κράτες που σέβονται, τις χώρες που σέβονται το κράτος δικαίου να οθήσουν τα δικά τους ε, συμφέροντα. Και θα πρέπει να εντάξουμε αυτά τα ζητήματα σε όλες τις σχέσεις μας με όλους τους εταίρους, τις τρίτες χώρες εταίρους. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Νομίζω και εγώ όπως όλοι ότι η έκθεση είναι περιεκτική, αναφέρει πολλά θέματα ασφάλειας και διεθνή συμφέροντα. Δεν αναφέρεται η σημασία της στρατηγικής διεύρυνσης σε σχέση με τη διαδικασία που άρχισε πριν από καιρό και που ακόμα λειτουργεί. Είναι ζωντανή. Εγώ θα υποβάλω, θα καταθέσω μια τροπολογία για τη διεύρυνση. Τα κεφάλαια για τις σχέσεις μας με την Ρωσία στην έκθεση είναι ισορροπημένα και με βρίσκουν σύμφωνο. Αλλά δεν είμαι βέβαιος για τη στρατηγική αν και κατά πόσο η στρατηγική των κυρώσεων ε, έδωσε θετικά αποτελέσματα. Φοβάμαι ότι ενίσχυσε το καθεστώς του Πούτιν και έβλαψε σοβαρά τα δικά μας οικονομικά συμφέροντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον Έλμαρ Μπρόκ, τον διακεκριμένο συνάδελφο και συγητή, για μία ακόμα καλή έκθεση και ιδιαίτερα για την παράγραφο 2. Το μέλλον της ε, ΚΕΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από το πώς θα αναγνωστεί αυτή η παράγραφος από τους διάφορους εμπλεκομένους. Ε, συμφωνούμε με την ε, ρεαλιστική διάγνωση και τους φιλόδοξους στόχους, όχι για πρώτη φορά, η ενισχύση των αμυντικών δυνατοτήτων μας θα γίνει πραγματικότητα αν υπάρξει το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο και η πολιτική βούληση. Αυτό το είπαν και άλλοι συνάδελφοι Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να συμμεριζόμεθα τις ίδιες απόψεις για τη Ρωσία, την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και άλλες εστίες, θερμές εστίες. Και αυτό μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί. Και είναι σαφές ότι η ήπια δύναμη δεν αρκεί. Τώρα η παράγραφος 29. Ε, θα προσέθετα και το διαπολιτισμικό διάλογο η πολιτιστική ε, διπλωματία αναφέρεται, αλλά νομίζω ότι δεν εξαντλούμε την ήπια δύναμη που υπάρχει εδώ. Τέλος, δεν νομίζω ότι όλοι οι εταίροι και οι περιφέρειες θα πρέπει να αναφερθούν, αλλά συμφωνώ με τον κύριο Βάγκλο ότι ε, τα Δυτικά Βαλγάνια πρέπει να αναφερθούν ειδικά και θα προσέθεται επίσης και την Ινδία και την Ιαπωνία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα μιλήσω ισπανικά, αλλά δεν θα διαφοροποιηθώ από το, του συναδέλφου. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ για την εξαιρετική έκθεση ε, ανωτά του επίπεδου που μας έχει συνηθίσει. Συμφωνώ λοιπόν με την έκθεση, πιστεύω ότι είναι πολύ ισορροπημένη και εστιάζει στα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ απόλυτα με τις παραγράφους 1 και 2, όπου αναφέρει τα θετικά της Ένωσης. Ίσως πρέπει να προσθέσουμε και την παγκοσμιοποίηση, γιατί νομίζω ότι εδώ ε, μιλάμε για κάτι που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Αναφέρεται ε, τις, ε, τα θετικά, τις αρετές της Ένωσης, ε, που συχνά ξεχνάμε. Στις, βέβαια δεν μπορούμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες στην έκθεση, αλλά πιστεύω ότι η παγκόσμια στρατηγική θα αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια, οπότε υπάρχουν αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο και είναι νομίζω πολύ σημαντικό να προχωρήσει η κοινή εξωτερική πολιτική μας και η πολιτική ασφάλειας. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα θετικά του Brexit. Δηλαδή θα επιτελέσουμε πρόοδο εδώ θα προχωρήσουμε σε τομείς όπου όπως ε, αναφέρθηκε η Πια δύναμη δεν αρκεί. Ε, στη Ρωσία, σε σχέση με τη Ρωσία, όπως και πολλοί άλλοι, πάντα ήμουν υπέρ της συνεργασίας, γιατί είναι σημαντικός ε, διεθνής παράγων, αλλά αυτά που γίνονται στη Συρία τώρα είναι πολύ απογοητευτικά. και δεν προϊονίζονται τίποτε καλό για τις μελλοντικες σχεσεις σχέσεις Ρωσίας-Ένωσης. Θέλω τώρα να αναφέρω δύο λεπτομέρειες. Ε, συμφωνώ απόλυτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύναμη μετασχηματιστική. Ε, αναφέρθηκαν ε, όλα αυτά και πώς βοήθησε και η διεύρυνση. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι στην παράγραφο 29 η νομοθετική ε, εξουσία είναι σαφής. Αναφέρεται η δύναμη της Ευρώπης, η κανονιστική. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το επεξεργαστούμε καλύτερα αυτό, να μιλήσουμε για το δικαιικό μας σύστημα. Τώρα, οι αναφορές στην ε, πολυμερή συνεργασία και διάσταση δεν έχει αναπτυχθεί πολύ. Μου φαίνεται ότι η έκθεση είναι πολύ καλή, αλλά θα ήθελα να ε, κάνω κάποια πρόταση για την παραγράφο 7. Μιλάτε για την άμυνα, ανάπτυξη και διπλωματία. Εγώ θα άλλαζα τη σειρά. Θα μίλαγα για διπλωματία, άμυνα και ανάπτυξη. Ή μάλλον διπλωματία, ανάπτυξη άμυνα. Ε, μου Δηλαδή διπλωματία, ανάπτυξη και άμυνα. Με αυτή τη σειρά πρέπει να αναφέρομαι τους τρεις αυτούς τομείς. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για το σχέδιο έκθεσης. Ε, έχουμε μεγάλες προσδοκίες γι' αυτό και δεν μας απογοητεύσατε. Είναι εξαιρετική η έκθεσή σας. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, αλλά φυσικά η συζήτησή μας ε, αφορά τον βελτίωση ακόμα περισσότερο αυτού του εγγράφου. Ελπίζω δηλαδή αυτή η έκθεση να αποτελέσει ένα σαφές βήμα προς τα εμπρός, ώστε να συμφωνήσουμε ε, για ποινίες Παγκόσμια στρατηγικής, όπως ε, ανέφερε η κυρία Μουγκερίνη. Ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλά θα υιοθετήσει μια παγκόσμια στρατηγική, αλλά θα αποτελέσει στρατηγικό παράγοντα σε παγκόσμια κλίμακα. Πράγματι, ε, έχετε κάποια καλά σημεία εδώ όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ κάτι απολύτως αναγκαίο δεδομένης της επισφαλούς ε, παγκόσμιας σημερινής κατάστασης. Αλλά να τονίσω συνεργασία όχι μόνο με το ΝΑΤΟ και διατλαντική συνεργασία και διατλαντική δεσμή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ χρειάζονται σε μεγάλο βαθμό. Όχι απλά να αφήνουμε τα πράγματα να πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση να πάρει σε κατεύθυνση μετά από τις προεδρικές εκλογές είπα, Ελπίζω αυτή η συνεργασία να παίξει σημαντικό ρόλο και για τις δύο πλευράς και να μην έχουμε απομονωτικές τάσει οποιοδήποτε είδους. Πραγματικά συμφωνώ με του συναδέλφου, οι οποίοι ανέφεραν τη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι ένα σημαντικό εργαλείο μεταρρυθμιστικό και για τη συνεργασία με τι γειτονές χώρε. Ταυτόχρονα στην παραγράφο 18 που αναφέρεται τη στενή συνεργασία με τους ανατολικούς εταίρους αυτή η παράγραφος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφής. Πρέπει να αφορά διμερείς δεσμεύσεις. Και εδώ πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε καθυστερήσει. Εμείς οι ίδιοι, οι χώρες αυτές έχουν καλές επιδόσεις. Έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο ε, με τη Συμφωνία Απαλλαγής θεωρήσει και εμεί έχουμε καθυστερήσει. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Ε, δεν μπορούμε να συμφωνούμε εδώ σε τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. και αυτή η καθυστέρηση είναι επιβλαβή και για τι δύο πλευρέ. Πρέπει, πιστεύω, να ε, παρέχουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί αφού έχει επιτευχθεί η αιρεσιμότητα. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι, να συμπεριλάβουμε κάτι γι' αυτό εδώ. Και τέλο, κύριε Πρόεδρε, Αργότερα σήμερα θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Φωτίγα για την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πραγματικότητα δεν είναι πάντα τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Υπάρχει πόλεμος πληροφοριών κατά τις δύση. Και το να το αναφέρατε στη δική σας έκθεση πιστεύω θα έκανε τα πράγματα καλύτερα και θα προσέδε μεγαλύτερη συνοχή γενικότερα. Γι' αυτό το λόγο ε, θα υποβάλουμε εμεί από πλευρά μα αυτέ τι τροπολογίε που θα υποβάλουμε και πάλι συγχαρητήρια για το σχέδιο εκθέση. Ευχαριστώ πολύ. Λέει Γκάλερ. Και εγώ επικροτώ την κατεύθυνση αυτής της έκθεσης και χαίρομαι για την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε την ε, διεθνή πραγματικότητα αλλά και τις συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν από τον Brexit. Θα ήθελα να σταθώ σημείο 10 και στις διάφορες παύλες που έχει το σημείο αυτό γιατί εκεί αναφέρεται το θέμα του γενικού στρατηγίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάπως σαν μια παράδοξη πρόταση πολλές ε, πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Η δημιουργία ενός ε, μόνιμου στρατιωτικοπολιτικού αρχηγείου με την ε, ολοκλήρωση των υπαρχόντων φορέων. Μα έχουμε ήδη στρατιωτικές ε, πολιτικές δομές, τα πάντα. Υπάρχουν όλες αυτές οι δομές. Το θέμα είναι πώς μπορούν να συνενωθούν αυτές για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα από ορισμένα κράτη-μέλη είναι ότι τους απασχολεί το θέμα της αποτελεσματικότητας αυτών των φορέων να συνενωθούν. Στα αγγλικά αυτό το οποίο διατυπώνεται δεν είναι μοναχά ο σχεδιασμός, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή και η δράση. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο σχεδιασμός στις Βρυξέλλες, αλλά η εφαρμογή των σχεδίων αφορούν τα κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Πρέπει να έχουμε planning and conduct στα αγγλικά, δηλαδή και η εκτέλεση των σχεδίων, όχι απλώς μονάχα ο σχεδιασμός. Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό αφορά τις αποστολές της ΚΕΠΑ και όχι κάτι άλλο. Ε, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταπραίνουμε τις ανησυχίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί από διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και κάτι ακόμα. Υπάρχει αυτό το οποίο λέγεται για την ε, πολιτική ε, άμυνας και ασφάλειας, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κινητοποιηθεί η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η ΠΕΣΚΟ. Θα έπρεπε να μπορούσαμε ήδη να έχουμε προχωρήσει στην υλοποίηση της ΠΕΣΚΟ. Μπορούν εκεί να συμμετάσχουν όλοι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται και μπορεί λοιπόν να υπάρξει στη συνέχεια μια ενσωμάτωση της, της δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ενωσιακές δομές μέσω του προπολογισμού που θα της δώσει πολύ μεγαλύτερη λειτουργικότητα και πολύ μεγαλύτερη ικανότητα να, αποτύχουμε, να επιτύχουμε τους στόχους μας. Για τις κυρώσεις τώρα, εγώ πιστεύω ακόμα ότι ήταν απαραίτητες και εξακολουθούν να είναι απαραίτητες ε, οι κυρώσεις και μετά από τις πρόσφατες ε, εξελίξεις στη Συρία θα πρέπει να ενισχυθούν. Αλλά δεν είναι το θέμα μονάχα αν έχουν αποτέλεσμα ή όχι. Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει πολιτισμένα τη δράση της Ρωσίας, αλλιώς θα έπρεπε να είχαμε στείλει στρατό και όπλα για να εξοπλίσουμε το, την Ουκρανική κυβέρνηση. Αυτό έκανε η Ρωσία από τη δική της πλευρά. Εμείς δεν ανταποδώσαμε τα ίσα. Απλώς Φέραμε αυτές τις ε, κυρώσεις με στόχο να πείσουμε τη Ρωσία να επανέλθει σε μια διπλωματική λύση για τα προβλήματα αυτά. Τώρα, από μια τέτοια στάση μέχρι το να φτάσουμε να πούμε ότι οι κυρώσει είχαν αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα, αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό να το πούμε. Εμεί αντιδράσαμε με πολιτισμένο τρόπο και όχι με τον ίδιο τρόπο που έδρασε ο επιτιθέμενο από τη ρωσική πλευρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φρόιντ, και εσείς ε, μαζί με τους ε, σοσιαλδημοκράτες θα θέλατε να προσθέσετε. Έχω το κείμενό μου στα αγγλικά και μπορώ να επανέλθω λοιπόν σε αυτή τη γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι λίγο άβολα, αλλά δεν θυμάμαι πότε πρόσφατα έχω δει τόσο μεγάλη υποστήριξη προς έναν εισηγητή και θα προσθέσω και εγώ τη δική μου υποστήριξη και τους επένους μου. Η μόνη επιφύλαξη αν μπορώ να την ονομάσω έτσι από αυτές τις συνθήκες, από πλευράς μου, είναι ότι όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα. Ίσως πριν από ένα χρόνο ή και παλιότερα. Και κάτι άλλο θα ήθελα να προσθέσω, που θα ήθελα έτσι να υπογραμμίζετε λίγο περισσότερο στην έκθεση, από ότι αυτή τη στιγμή είναι η Συρία και η απόλυτη μας αδράνεια μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε καταφέρει να καλύψουμε το κενό που έχει διαμορφωθεί μετά από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και είπα ΕΕ. Είναι κάτι που ουσιαστικά αποτελεί έκκληση βοήθειας ε, προς την Ευρώπη για να βοηθήσουμε τα 500 εκατομμύρια πολίτες που, που μας εκλυπαρούν για επίλυση αυτής της ε, σύραξης. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, πιστεύω. Ειδικότερα δεδομένου των συνθήκων, δεδομένου του πόσο μας επηρεάζει αυτή η σύραξη, περισσότερο από ό,τι κάθε άλλη σύραξη στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα σας επενέσω όπως και οι υπόλοιποι. Κύριε Μπρόκ, ε, έχετε συντάξει ένα εξαιρετικό σχέδιο έκθεση που επισημαίνει όλα τα σημαντικά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη εξωτερική πολιτική τη. Συμφωνώ με το μήνυμα που δίνεται ότι η σημερινή κατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για τη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Επίσης διαβάζω στην έκθεση ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις θετικές πτυχές της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής όπως το συνεργατικό μας πνεύμα στο διεθνές στερέωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τη σχέση της με τους στρατηγικούς εταίρους και να παραμείνει αξιόπιστος ε, παράγοντας την παγκοσμία σκηνή. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είναι ενωμένη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες ε, στη διεθνή σκηνή, όπως για παράδειγμα στα Ηνωμένα Έθνη. Κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, καθόλου μάλιστα. Επίσης πιστεύω πρέπει να εστιαστούμε και στη γειτονία μας, να αξιολογήσουμε τους στόχους και τα επιτέγματά μας εκεί. Και πρέπει να δούμε ότι τα εργαλεία εξωτερικής μας πολιτικής λειτουργούν και επηρεάζουν θετικά την εξωτερική πολιτική. Όσον αφορά την ασφάλεια, πρέπει να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για κάτι περίπλοκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολλέ απειλέ για την ασφάλεια. Την τρομοκρατία, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ασφάλεια των εξωτερικών μα νόρων, την ενεργειακή ασφάλεια και ούτω καθεξή. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί ενισχυμένη συνεργασία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με του παγκόσμιου εταίρου και οργανισμού μα. Τι θα κάνουμε με την έκθεση τώρα, Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι καλό θα ήταν να προσθεθούν προτάσεις εδώ και εκεί ώστε να τονίσουμε τα σημαντικά σημεία της μελλοντικής στρατηγικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται κάποιο ε, δούλεμα λεπτομέρειες, αλλά με τρόπο τέτοιο που να μην ε, ε, χαλάσει την ισορροπία που επιτυγχάνεται σε αυτή την εκθέση λόγω της πολύπλοκης φύσης της. Αυτό πιστεύω είναι το κλειδί. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για όλες σας τις ε, καλές ε, παρατηρήσεις. Also, einmal... Λοιπόν, για να δούμε. Του ε, ρώτησε η Καλνιέτη για τα 2%. Τα 2% αύξηση των αμυντικών δαπανών δηλαδή αύξηση στα 2%, ε, έχει την αξιοπιστία το 0,7% για τους στόχους της χιλιετίας. Πόσο ε, συχνά το είδαμε να πραγματοποιείται. Έτσι είναι, ρεαλιστές να είμαστε. Και αν δούμε το, την κατάσταση σήμερα, οι συνέργειες νομίζω ότι δίνουν περισσότερα αποτελέσματα. Δεν αποκλείω το 2%, αλλά μου φαίνεται ότι με τις συνέργειες θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μπορούμε να έχουμε και 200 δις ε, για την άμυνα. Κάποια κράτη-μέλη έχουν 80% ή μέχρι 80% γενικά έξω, θα δαπάνες σε αυτό το τομέα. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν να καλυφθούν οι ανάγκες των στρατιωτών. Και 46-48% είναι οι γενικές δαπάνες και στη χώρα μου, στη Γερμανία. Δηλαδή οποιαδήποτε επιχείρηση θα επιτόχευε. Έχουμε λιγότερους στρατιώτες, αλλά έχουμε τους ίδιους διοικητικούς υπαλλήλους. Μου φαίνεται ότι το ίδιο συμβαίνει ε, ε, παντού. Δεν μειώθηκε ο διοικητικός μηχανισμός ε, πριν από λίγα χρόνια, αλλά μειώθηκε ο αριθμός των ενόπλων. Η συνέργεια είναι κάτι που πρέπει να το κοινοποιήσουμε. Αυτό που κάνουμε σήμερα, αυτό που κάνουν το κράτη-μέλη, λόγω της άρνησης συνεργασίας, εκεί όπου ε, εξοικονομούνται δαπάνες ε, είναι ο τομέας της ε, έρευνας, των προμηθειών. Αυτό είναι αποφασιστικός παράγον και εκεί μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερη χρήση για τα χρήματά τους από ό,τι μέχρι τώρα. Δηλαδή πρέπει η συζήτηση αυτή να γίνει δημόσια γιατί Υπουργοί Άμυνα δεν θα κάνουν δημόσια συζήτηση. Θα συζητήσουν μόνο για θέματα εθνικής κυριαρχίας. Όταν όμως γίνει συζήτηση και στο τομέα του, της άμυνας, θα πρέπει να εντάξουμε και τους ε, υπουργούς στη συζήτηση αυτή. Πολλοί μίλησαν για το κέντρο διοίκησης ε, ή το αρχηγείο. Νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό το θέμα, να έχουμε ξεκάθαρες απόψεις. Αναφέρθηκαν σχετικές προτάσεις. Ενδεχομένως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν μια συνάντηση για να συζητήσουν το θέμα αυτό και να καταλήξουν σε μια ωραία συμβιβαστική τροπολογία. Ομίζω, ο κύριος ε, Κούκαν, κύριε Κούκαν, το θέμα του fine tuning και το θέμα της ενημέρωσης στο θέμα Συρία θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, να κάνουμε τη σχετική ενημέρωση γιατί τέλειωσα ε, όταν ακόμα δεν είχα καταλήξει ε, σε σχέση με το θέμα της Συρίας, δεν είχα δηλαδή τις απόψεις που έχω τώρα. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια ενημέρωση. Τώρα, το δύναμη ήπια και σκληρή Εμείς νομίζω ότι πρέπει να το θέσουμε ως εξή ότι πάντα θέλουμε να προλαμβάνουμε τις συγκρούσεις. Όλα τα άλλα συνιστούν πολιτική αποτυχία καμιά φορά. Χρειάζεται βέβαια και σκληρή βία για την αποτροπή της σύγκρουσης. Και αυτό δεν το παρέχουμε. Είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές, χρηματοδότες και θα είμαστε και στην ανοικοδόμησή της οι μεγαλύτεροι δωρητές, αλλά κανείς δεν μας παίρνει στα σοβαρά όταν πρόκειται για πόλεμο και ειρήνη. Είναι σημαντικό αυτό να μας πάρουν στα σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα κέριο που πρέπει να το λύσουμε για να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Για τη διεύρυνση τώρα ο κ. Φάιγκλ. Θα δούμε πώς θα το συνδέσουμε αυτό. Είπαμε ότι η διεύρυνση είναι σημαντικός πολιτικός στόχος και η μέχρι τούδε διεύρυνση ε, ήταν ένας στόχος εξωτερικής πολιτικής ε, ειρηνευτικός, έγινε αυτό, αλλά η διεύρυνση έχει και όρια. Δεν είναι αέναη, θα πρέπει να ε, συνάδει με την λειτουργική ικανότητα της Ένωσης και ίσως πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ πλήρους ένταξης και της σημερινής κατάστασης με μηχανισμούς όπου μπορούμε να έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο συν να προσφέρουμε δηλαδή κάτι προσελκύοντας πιο κοντά μας τις χώρες, γνωρίζοντας όμως ότι ε, που δεν είδε πληρούν τους όρους για πλήρη ένταξη, αλλά ούτε και εμείς δεν μπορούμε να ε, λειτουργήσουμε ε, αν υπάρξουν ανεξέλεγκτες προσχωρήσεις. Ε, σε αυτό δεν θέλω να με ε, παρεξηγήσετε. Με τα νέα δεδομένα χρειάζεται ένας νέος μηχανισμός. Ενδεχομένως, σημαντικότερο να είναι αυτό για τις χώρες της ανατολικής πολιτικής γειτονίας, ίσως και για την Τουρκία αν έχετε βελτιωτικές προτάσεις για να γίνει πιο αυστηρό το κείμενο και πιο ξεκάθαρο, ευχαρίστως. Θα είμαι ευγνώμων. Και αυτό ισχύει και για τον κύριο Πέτερλε. Για την παγκοσμιοποίηση. Να δούμε τι ακριβώς πρόβλημα έχετε, γιατί δεν κατάλαβα περί τίνος, πρόκειται. Για το Brexit, Είναι σαφές ότι η Βρετανική αποχώρηση συνεπάγεται αποδυνάμωση της ικανότητάς μας και στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα. Ε, με όλες τις δυνατότητες που έχουμε μετά την αποχώρηση. Το καλύτερο ε, θα ήταν να έχουμε ενταγμένη με επικοδομητικό τρόπο τη Βρετανία στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας αν συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις μετά, για τον Brexit, θα πρέπει να γίνουν και αναφορές ε, στις ε, μελλοντικές ικανότητες στους τομείς αυτούς της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν μπορούμε να τα αποσυνδέσουμε όλα αυτά και ίσως θα, ε, θα, θα, υπάρξουν ιδέες και προτάσεις για το πώς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα με τη Βρετανία. Δεν μπορεί να τη θεωρήσουμε δηλαδή έτσι απλά τρίτη χώρα. Τώρα, για τις κανονιστικές εξουσίες, ενώ διεθνές δίκαιο, αλλά και τα θέματα πολιτιστικής συνεργασίας. Μπορούμε να το διατυπώσουμε καλύτερα για να αποφευχθούν οι παρανοήσεις. Ε, βεβαίως, διπλωματία, ανάπτυξη, άμυνα. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Ο συνάδελφος Αστρεβίτσιους το ΝΑΤΟ για την Ευρώπη είναι απολύτως αναγκαίο για τη συλλογική ασφάλεια. Και αυτό το λέμε. Αλλά λέμε και πέραν τούτου ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες με την Αμερική πρέπει να ενισχυθούν. Αν βρείτε πρόταση άλλη η οποία θα βρει σύμφωνο όλο το Κοινοβούλιο θα ήμουν ευγνώμων. Αλλά δεν θα ήθελα στην έκθεση αυτή να προχωρήσω σε αντιπαράθεση εις ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και μέχρι ποιου σημείου πρέπει αυτές να προχωρήσουν. Θέλουμε συνένεση, θέλουμε να αποφύγουμε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Στο Κοινοβούλιο μου φαίνεται ότι γίνομαι κατανοητός. Τώρα, οι διαδικασίες για τις θεωρήσεις, δεν θέλω να το πω αυτό γιατί πρέπει μάλλον να έχει τελειώσει μέχρι το Δεκέμβρη, οπότε θα είναι ήδη ξεπερασμένο. Τι έγινε με το τι έκβαση είχαν οι συζητήσεις στο τριμερή διάλογο. Δεν πήγανε καλά. Ε, πέρα από την ε, έκθεση μου, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα και προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου θα πρέπει να μιλήσουμε και για το θέμα της εφαρμογής εκτέλεσης ε, των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Κοινοβουλίου, αλλά ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε και την λειτουργική δράση μας, την λειτουργικότητα. Ε, δεν μπορεί να είναι μόνο το κοινοβούλιο λογικό, πρέπει να είναι και η Κομισιόν και το Συμβούλιο, γιατί το Συμβούλιο λέει να είσαστε λογικοί. Αυτό μπορώ να το αντιστρέψω για να ισχύσει και απέναντι στο Συμβούλιο αυτό, αυτή η παρένεση. Δεν είναι καλό τους ε, εκπροσώπους του Συμβουλίου της Γεωργίας, της Ουκρανίας ε, να τους ε, λέμε ότι το Κοινοβούλιο δεν υποχωρεί. Είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να το παίζει το Συμβούλιο και κάποια στιγμή θα πρέπει να το καταλάβει το Συμβούλιο και να προχωρήσει σε βελτιωμένη διαδικασία. Τώρα για τα κεντρικά, κεντρική διοίκηση το αρχηγείο, ε, νομίζω ότι είπαμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό ε, και το σχεδιασμό και τη διενέργεια ή την εφαρμογή ικανοτήτων. Ε, και, και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ε, Πρέπει να το αναλύσουμε αυτό ε, το θέμα, δεν είναι μόνο μια σύνοψη. Θα πρέπει να δούμε ε, και την προστιθέμενη αξία που θα σημάνει ένα ποιοτικό άλμα. Αυτό το ποιοτικό άλμα θα πρέπει να το αναδείξουμε περισσότερο, ούτως ώστε να φανεί, να καταστήσουμε σαφή τη διαφορά. Μου φαίνεται ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω από σας τώρα τις ε, τροπολογίες και αν υπάρξουν και τίποτε, αν, υπάρχουν παρανοήσεις, ευχαρίστως να τα ε, συνεννοηθούμε όλα αυτά και να τα ρυθμίσουμε. Εντάξει, τελειώσαμε. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έρχομαι όμως τώρα στην πιο σημαντική έκθεση. Εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία πλευρά και της Κολομβίας και του Περού από την άλλη μεριά για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Εκουαδόρ. Εδώ έχουμε μία κάπως τεχνικού χαρακτήρα έκθεση αλλά, και δεν θέλω να κάνω μία παρουσίαση αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήματα που θέλετε θέση. Εάν δεν υπάρχουν ούτε ερωτήματα, να σας αναφέρω το χρονοδιάγραμμα. 4 Οκτωβρίου έχει εκπνεύσει η προθεσμία για τις τροπολογίες. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε για τις τροπολογίες, αν τις έχουμε βέβαια. Α, μα δεν υπήρξαν τροπολογίες καθόλου, λέει η γραμματεία. Στις 12 Οκτωβρίου λοιπόν θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ο κύριος Χάουιτ όμως προηγουμένως. Πραγματικά δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μια από τις τελευταίες μου αρμοδιότητες ε, ως, ε, στην Επιτροπή αυτή θα είναι μια σχέδια συζήτηση, οπότε να πω δύο λόγια. Ανέκαθεν προσπαθούσαμε να ασχοληθούμε με την περιοχή του σημερινού και εκείνη την περιοχή. Πιστεύω ότι η συμμετοχή του είναι κάτι καλό και για την περιοχή και για εμάς. Περιβαλλοντικά είναι πολύ ευαίσθητο το μέρος αυτό λόγω των οικοτόπων που υπάρχουν. Είναι από τα βασικά σημεία βιοπικιλότητας στον κόσμο, οπότε καλό είναι να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Εγώ έχω ασχοληθεί προσωπικά με συναδέλφους από τον Ισημερινό και ειδικότερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνθήκης για τα άτομα με αναπηρία και ο Ισημερινός είναι μια από τις χώρες που βοήθησαν και τους είμαι ευγνώμων γι' αυτός. Επίσης είναι ένα από τους κυρίους στο σύστημα του των Ηνωμένων Εθνών για ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ένα λυπηρό ιστορικό, αλλά προσπαθούν να το αναστρέψουν, να το αντιστρέψουν, συγγνώμη. Και φυσικά έχουμε και τον πρέσβη του Ισημερινού από τη Γενέβη εδώ στις Βρυξέλλες, οπότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε προσωπικά, οικονομικά, είναι κάτι πολύ καλό είναι μια γνωμοδοσία για την Επιτροπή Ήτρε και συμφωνώ με τα όσα είπατε. Πρέπει να μην ξεχνάμε τη σπουδαιότητα τη πολιτική συνεργασία μεταξύ ημών και του σημερινού. Και καλωσορίζω τι συστάσει προ την Επιτροπή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε λιγότερα από αυτά που κάνουν άλλες χώρες. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του τύπου είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί στην έκθεση με τον καταλληλότερο τρόπο. Δεν ξέρω ο κύριος Σόλτς έχει την πρόθεση να διατυπώσει ένα ψήφισμα για όλα αυτά. Ο κύριος Σόλτς είναι πάντα έτοιμος να αναφερθεί σε άλλες χώρες αλλά όχι στο Εκουαδόρ. Ενδεχομένω να υπάρξει ενδιαφέρον λοιπόν για ένα τέτοιο ψήφισμα. Εάν θέλει λοιπόν σε λίγες προτάσεις να πει ότι θέλουμε λοιπόν την συνεργασία αλλά με κάποιες ε, προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει λόγο. Όχι. Ich glaube, wir sollten, haben wir... Αύριο έχουμε την ε, συζήτηση για την Κολομβία στην Μέση Δίδαξη και τη Γεωργία επίση. Έχουμε διάλειμμα τώρα μισή ώρα μέχρι τι ε, ψηφοφορίε. λέει ο πρόεδρος. Δεν ξέρω, μάλλον έχουμε μισή ώρα, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο επίκαιρο θέμα που θέλετε να συζητήσουμε σε αυτό το διάμεσο διάστημα. Θέλετε να πούμε κάτι για τη Συρία. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, αν θέλετε Συρία, Συρία. Αν θέλετε διακοπή, διακοπή. Γιατί βλέπουμε ότι οι αντιπαραθέσεις οι οποίες έχουν ε, λάβει χώρα τα τις τελευταίες μέρες μας οδηγούν σε μεγάλες δυσκολίες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δούμε πώς μπορεί να εξευρεθεί μια λύση μεταξύ και Ηνωμένων Πολιτειών και της ε, Ρωσίας για να υπάρξει μια ανακοχή η οποία θα ενισχύσει την διαδικασία ειρήνευσης στη Γενέβη. Είχε γίνει προσπάθεια προσέγγισης με την κυβέρνηση του κυρίου Ασάντ, αλλά τα γεγονότα τώρα δείχνουν ότι δεν είναι πρόθεση η προσέγγιση, αλλά η επίτευξη μιας λύσης μέσω στρατιωτικών μέσων. Η προσφορά να εγκαταλείψουν όσοι θέλουν το χαλέπι αυτή τη στιγμή, αυτό σημαίνει τους καλεί να αποδεχτούν μια ήττα και να υποταγούν και πάλι στην κυβέρνηση του Ασάντ. Δεν μπορεί κανείς, πώς μπορεί κανείς σε, μακροχρόνιο επίπεδο να αφήσουμε να ηγείται μιας χώρας στην οποία αυτός πολεμάει τον ίδιο του τον λαό, τον ίδιο τον λαό του χρησιμοποιώντας ακραία βία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαπιστώσουμε και για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία των διαπραγματεύσεων της ε, Γενέβης όπου είναι όλοι παρόντες, ακόμα και οι χώρες που κάνουν πόλεμο δι αντιπροσώπων από τη Σαουδική Αραβία μέχρι το Ιράν, η Τουρκία, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να βρούμε μια συμφωνία που θα μας επιτρέψει να στραφούμε όλοι μαζί κατά του Ισλαμικού κράτους. Αυτή η πολιτική θα μειώσει την προσβηγική ροή θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναγυρίσουν στις αιστείες τους και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να μπορέσουμε να επαναφέρουμε μια λογική κρατική δομή στη Συρία εάν ο μόνος τρόπος να βρεθεί μια λύση είναι η βία Υπάρχει ο κίνδυνος γενικού κατακαιρματισμού στην ε, περιοχή. Τι θα γίνει με, την, ε, με τις τρεις κουρδικές ενότητες και την εδαφική αικαιρεότητα της Τουρκίας και της Συρίας που συνδέεται με αυτό το πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν υπάρξει η λύση με την ήττα του Ισλαμικού κράτους κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε μια τελείως διαφορετική διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης στην περιοχή αυτή. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποδεχτούμε, αλλά ξέρουμε όλοι ότι μια δημοκρατική οντότητα όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε ή η Ευρώπη έχουν λιγότερες δυνατότητες αντίδρασης σε μια τέτοια κατάσταση από ότι ένα αυταρχικό κράτος όπως ε, η Ρωσία. Πρέπει λοιπόν να βγούμε από το καλούπι της σκέψης που έχουμε μέχρι και να ξανασκεφτούμε από την αρχή για όλα αυτά τα θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει στο παρελθόν ήταν λάθη. Σε προηγούμενες χρονικές στιγμές, όταν έγινε η δημοκρατική εξέγερση στη Συρία, ήταν σωστό να την υποστηρίξουμε. Αλλά για όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε και κάποια δυνατότητα αυτοκριτικής. Ίσως ήταν σφάλμα το ότι μπήκαμε στη Λιβύη, αλλά δεν μπήκαμε, ενώ δεν μπήκαμε στη Συρία. Δεν είχαμε επέμβαση στρατιωτική στη Συρία. Αλλά από την άλλη πλευρά λένε πάρα πολύ ότι η Ευρώπη απέτυχε στη Συρία. Μα εμείς δώσαμε μονάχα ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Μα τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει. Ποιος θα ήταν έτοιμος να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Συρία. Και είναι εύκολο να θέτουμε το ερώτημα, αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος είναι διατεθειμένος να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε μια χώρα όπως η Συρία. Έχουμε την ανάγκη να δούμε τα πράγματα όχι με έναν τρόπο ο οποίος επιρρύπτει την ευθύνη για την αδράνεια στην Ευρώπη, αλλά όχι στα κράτη-μέλη Αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή καμία απάντηση σε αυτό το ερώτημα του πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Φρόντ, ούτε και απάντηση. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Ε, είναι εύκολο εκ των υστέρων να λες ότι δεν θα έπρεπε να επέμβουμε στη Λιβύη ενώ θα έπρεπε να έχουμε επέμβει στη Συρία. Προχύθηκε το γάλα. Είναι αργά. Είναι πολύ αργά. Πάντως δεν είμαστε και τόσο αδύναμοι όπως είπατε, όπως μας τα ε, παρουσιάσατε. Και δεν εννοώ τώρα τη στρατιωτική δύναμη, αλλά ένα άλλο επίπεδο. Αν έχουμε υπόψη μας ε, αυτοί που το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, τη Ρωσία, για να αναφέρω κάποιους από αυτούς που κάνουν πόλεμο δια αντιπροσώπου, Έχουμε πολύ στενές οικονομικές σχέσεις με ορισμένες από αυτές τις χώρες. Οι Γερμανοί έχουν ε, παραδώσει στρατιωτικό υλικό στη Σαουδική Αραβία της τάξεως αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ή δολαρίων. Έχουμε στενές οικονομικές σχέσεις και σχεδιάζουμε κι άλλες οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, οικονομικές διασυνδέσεις. Δηλαδή υπάρχει δύναμη από την πλευρά μας, έχουμε ένα μοχλό Με το οικονομικό μας βάρος μπορούμε να ασκήσουμε πίεση σε αυτές τις χώρες και να τους πούμε ότι αν κάποια δεν σταματήσετε επιτέλους τον πόλεμο τότε δεν θα σας δώσουμε ούτε έρμπας, ούτε αεροπλανοφόρα, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλα όπλα ε, παίρνει η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά τέρμα. Βέβαια μπορεί να πάνε και να τα αγοράσουν από άλλους, αλλά ίσως και εκεί να βρούμε συμμάχους που και αυτοί θα αρνηθούν. Ο Συριακός λαός ε, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να τερματιστεί ο πόλεμος εκεί και όχι μόνο να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και να λέμε τα δοκιμάσαμε όλα και δεν γίνεται τίποτε. Ε, ε, δηλαδή έχουμε στη φαρέτρα μας όπλα για να ασκήσουμε πίεση και επανέρχομαι σε αυτό που είπα και προηγουμένως ότι αυτό το κενό από το τερματισμό της ε, συνεργασίας Ρωσίας-ΙΠΑ για την ειρήνευση στη Συρία, αυτό το κένο ε, μπορούμε και πρέπει να το καλύψουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε τη συζήτηση αυτή με ερωτήσεις με ερωτήματα τα οποία είναι θέματα ουσίας και τα οποία δεν έχουν κατά ανάγκη κάποια σαφή απάντηση. Αλλά δεν είμαι σίγουροι ότι τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Αν δούμε την κατάσταση, έχουμε αυτή τη στιγμή μια συσσόρευση εμφυλίων πολέμων στη Συρία που κάνουν την κατάσταση όλο και πιο πολύπλοκη και επεπλεγμένη. Έχουμε μια μεγάλη δύναμη, τη Ρωσία, που έχει μια σαφή στρατηγική από ό,τι φαίνεται να συνεχίσει την κατάκτηση εδάφους προτού φτάσουμε σε διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση και συγχρόνως βλέπω ότι ενώπιον της Ρωσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άοπλη, δεν έχει μια στατηγική, δεν έχει μια σαφή προοπτική, ένα σαφές όραμα για το τι θέλει. Προφανώς υπάρχουν χώρες όπως η Δική Αραβία και το Ιράν, όπως είπε ο προλαλής σας, με τις οποίες όχι μόνο μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά μπορούμε να ασκήσουμε και κάποια πίεση. Βλέπουμε ότι η διάσταση περιφερειακού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντική στην περιοχή. Δεν μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία ειρήνευσης εάν δεν λάβουμε υπόψη τις, τα συμφέροντα αυτών των περιφερειακών δυνάμεων, ακόμα και αν είναι σε αντιπαράθεση μεταξύ τους αυτά τα συμφέροντα. Πολλές φορές μιλάμε για αυτή την ασφαλή ζώνη, μια προστατευμένη ζώνη, όπου μπορούν να ζήσουν εν ειρήνη οι πολίτες της Συρίας. Αυτό είναι μια πραγματική ουτοπία, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο εμείς ως Ευρωπαίοι μπορούμε να το ζητήσουμε, να το εξασφαλίσουμε. Αυτά το οποίο γίνεται σήμερα στο Χαλέπι και το προσφυγικό ρεύμα που έχουμε αντιμετωπίσει, τα 5 εκατομμύρια άτομα που έχουν φύγει από τη Συρία, όλα αυτά θα συνεχιστούν. Υπάρχουν εκατομμύρια εκτοπισμένων, εκατομμύρια ανθρώπων που πλήττονται από μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, νομίζω ότι η Ευρώπη έχει την υποχρέωση, τουλάχιστον ακόμα και αν δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις, να έχουμε μια στρατηγική και ίσως να προωθήσουμε την ιδέα των ασφαλών ζώων. Σας το λέω αυτό με κάθε ταπεινοφροσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Ποιος θα τσεγγιθεί αυτές τις ασφαλείς ζώνες, λέει ο πρόεδρος Μπροκ. Δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συμφωνία από όλους για να γίνει κάτι τέτοιο. Η Ρωσία προβάλλει πάντα ένα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και μα ξέρουμε ότι η Ρωσία έχει εγκαταστήσει και πυράβλους εδάφους αέρος δεν θα μπορούν τα αμερικανικά ή τα τουρκικά αεροσκάφη να εξασφαλίσουν την ασφάλεια αυτής της, ε, της ε, ασφαλούς ζώνης. Δεν μπορούμε πια να έχουμε μια ζώνη μη υπέρπτυσης. Γιατί τα αεροσκάφη τα οποία θα επεκτεύαν αυτή τη ζώνη κινδυνεύουν να βληθούν από πυράβλους εδάφους αέρος. Και επίσης είναι πολύ πιθανό να έχουν και οι αντιπολιτευόμενοι, οι αντάρτες μάλλον, οι δυνάμεις αντιπολίτευσης στην ε, Συρία πυράβλους εδάφους αέρος. Αυτό το είδαμε και στο Αφγανιστάν να γίνεται. Αλλά ίσως είναι και ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να καταρρύπτουν τα αεροπλάνα του Ασάντ. Αλλά ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει, είναι πια πολύ αργά. Επομένως δεν μπορεί να εξασφαλίσει σε στατικό, επίπεδο κάτι τέτοιο η Δύση αυτή τη στιγμή. Είδαμε αυτά που έγιναν τις τελευταίες 14 μέρες. Μπορεί να ακούγομαι πολύ απεσιόδοξος. Ναι. Αλλά ο κύβος ερήφθη και δεν είναι εύκολο να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Ωραία, σε 15 λεπτά θα αρχίσουμε την ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε. Ξαναρχίζουμε και πάμε στις ψηφοφορίες. Το σημείο 7. Η κυρία Φωτίγκα είναι η συγγήτρια. Δεν ήρθε. Α, δεν ήρθε. Ποιο θα την ε, εκπροσωπήσει ο κύριος Στάνοκ, ο Τσάρλς, η κυρία Φωτίδα για προσωπικούς ε, λόγους δεν μπόρεσε να έρθει και ζητεί συγγνώμη. Καλώς, συμβαίνουν αυτά. Ευχαριστώ. Ε, τροπολογία 103. πέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Ε, δεν ψηφίσατε τότε, γιατί αυτοί που ψήφισαν περισσότερο ήταν 122, ε, 121, ποιος είναι υπέρ. Κατά. έλεγχος. Πέρας. 17 υπέρ 18 κατά απορρίπτεται. Ε, και 18-18 να είναι. Πάλι απορρίπτεται. Καλή προσπάθεια. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τώρα. 136 υπέρ. Κατά έλεγχος. Πέρας. 21 υπέρ 22 κατά απορρίπτεται. Λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 149 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 153-154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας.

Απορρίπτεται. Ε, κατά είναι. Ε, είναι και άλλοι πέντε. Δεν νομίζω ότι είναι το ε, σύνηθες αυτό. Να φέρνετε την κάρτα σας. Αλλιώς μπορεί να μην μετρήσει η ψήφο σας. Συμβαστική 9. Α, όχι, όχι, όχι. 158, συγγνώμη. 158 γκάλερ. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρασε. 25 προς 20. Δεκτή. Πώς θα κάνουμε νέα προπαγάνδα άμα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα θέματα. 159. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρασε 27 προς 20. Δεκτή. Έχουμε αναπτυξιακή διαδικασία τώρα στο μυαλό από ό,τι φαίνεται των συναδέλφων από το ΕΛΚ. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά δεκτή. 184. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 186 υπέρ κατά αποχές δεκτή 187 υπέρ κατά αποχές δεκτή 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 190 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 215. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έλεγχος. Πέρας. Σωστό. Απορρίπτεται. 23 υπέρ, 26 κατά, 234 Πλένκοβιτς υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 235 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 236 υπέρ. Κατά αποχές δεκτής Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 συμβαστική υπέρ. Περ, κατά αποχές δεκτή. 249 ε, υπέρ. Όχι. Λάθος θα λέει ο κατάλογος. Ε, συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά ποχές δεκτή. ...265 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα... ...266 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ κατά έλεγχος. ...267. Πέρας. απορρίπτεται. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 269 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 271 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 274 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή όχι, όχι 280, όχι 200, 289 ε, υπέρ, κατά. Όχι, ο κατάλογος είναι λάθος. Είχα δίκιο λοιπόν. Α, λάθος με συμβούλεψαν λοιπόν. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές. Φαίνεται ότι απερίφθη. Ακαταπίπτει τελικά η 289. Η 289 καταπίπτει γιατί είχε γίνει δεκτή η τροπολογία 149. Πάμε τώρα στη 293 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστή 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 308. Πού είναι η 308 τώρα. Υπέρ. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 309 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ κατά αποχέ πάλι 310 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 311 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 322 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Το πρώτο τμήμα ε, ο πρόεδρος Μπροκ. Δεύτερο τμήμα να χαψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά. ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Άρχισε. Η Πέρας. 17.33 απορρίφθηκε. Παρακαλώ τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην ψηφοφορία, γιατί δεν μπορώ να, να εκτιμήσω αλλιώς το αποτέλεσμα σύμβαση και 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.30 υπέρ υπέρ 330 κατά αποχές εγκρίνεται 3.31 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Πέρας. 2031 απερίφθη. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3,55, υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 13 με 27 απορρίπτεται. 356 <clears throat> υπέρ. Οι σοσιαλιστές ψηφίσουν ναι στις, στις ε, ψηφοφορίες διαντάσεως χειρών και όχι στις ε, ηλεκτρονικές. Αυτή είναι μια δυτή στρατηγική. 356 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 357 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 358 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές 63 υπέρ λέγω κατά εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 67 μέχρι 69 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές τώρα μπερδεύτηκα τελείως λέει ο πρόεδρος 70 έλεγχο, όπω ζήτησε κάποιο ηλικιωμένο κύριο ε, στη μέση αίθουσα. Πέρα τη φοφορία. Με 34-13 εγκρίνονται. Ο κύριο Σαφχάζο με την 70 έχει τύχει λοιπόν. 71 λέει ο πρόεδρος, όχι εκπίπτει, όλες εκπίπτουν, όλες εκπίπτουν μέχρι κάτω, μέχρι κάτω, μέχρι τον κύριο 78 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 5 υπέρ, τι λέτε, η 79 εγκρίθηκε λέει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 95. Υπέρ. Κατά αποχές. Πάλι, πάλι. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος Die 25 25-27 απέριπτε. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος 25-27. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ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 κατά αποχές δεκτή, 16 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ, κατά αποχές Αν έχει ψηφίσει και για τον έχει, για το όχι, αλλά και για τις αποχές, λέξει στην κυρία Γκόμης ο πρόεδρος. 20 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αλλά νομίζω ότι εγκρίνεται. Άψιμο της Πέρας ψηφοφορίας. 31-18 εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτούρα 1 υπέρ κατά αποχές κουλτ 1 υπέρ κατά αποχές δεχτεί κουλτούρα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κουλτούρα 5 υπέρ κατά έλεγχος. Πέρασε. Εγκρίνεται 26-22. Κουλτούρα 6. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 7 υπέρ. Κατά αποχές 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις υπόλοιπες αφού έχουμε την ίδια πλειοψηφία κάθε φορά. Ορίστε. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή.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 «31 υπέρ, 8 κατά, 14 αποχές γίνεται δεκτή». Συγχαρητήρια. Προχωρούμε τώρα στην έκθεση Παντσέρη. για τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας, σχέδιο γνωμοδότησης. Θέλει να πει κάτι ο Δεν είναι εδώ. Απλουστεύονται τα πράγματα. Κυρία Γκίλ, θέλετε να μας πείτε πολλά? Όχι. Συμβιβαστική ένα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 20. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 21. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τώρα, η τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή, Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται, 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ε, τροπολογία 73, όχι, έχει αποσυρθεί. Η 74, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 76 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 77 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, Ναι, ελεύθερη ε, ψηφοφορία 10. Όχι, όχι, όχι. Ε, την 9 υπέρ. Συμβαστική 9. Κατά αποχές δεκτή. Τώρα συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 90 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 91 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 92 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 93 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 94 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 95 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, ε, όχι, καταπίπτει 96. 1 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή, 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. Πέρα. 46 υπέρ. Δύο κατά δύο αποχές. Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ένας ε, μεταξύ των δύο ψήφων κατά. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Και νομίζω τελειώσαμε. Αύριο θα αρχίσουμε το πρωί 9 και 30. 9 και 30 αύριο. Auch missverständlich. <laughs> ja. Wünsche schönen Abend. Καλό σας βράδυ.